Right, Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε που καθυστέρησα λίγο. προσπαθήσαμε να βάλουμε και τη συνεδρία, την έναρξη της συνεδρίας λίγο πιο αργά από ό,τι κανονικά, αλλά φαίνεται ότι δεν πρόλαβα να έρθουν όλοι. Ε, εν περιπτώσει, στην ημερήσια μας διάταξη έχουμε τώρα να εξετάσουμε τις τροπολογίες για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων των δημοσιονομικών μέτρων για την ε, ανάταξη της οικονομίας. 162 τροπολογίες και θα παρακαλέσω τον ε, συνάδελφο Χουάν Γκόν να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. και επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστώ τους σκιώδεις ηγητές για την ε, συνεργασία τους. 162 τροπολογίες, πολύ επικοδομητικές επί της ουσίας. Είχαμε μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια συζήτηση που σε τελευταία ανάλυση κοινή και τους οικονομολόγους όλου του κόσμου όπως και τα μέλη της Επιτροπής μας. Και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η έκθεση και ο διάλογος τον οποίο ανέπτυξα με τους σκιώδεις συζητητές εντάσσονται σε ένα πνεύμα συμβιβαστικό, με αυτό το πνεύμα δηλαδή συνέταξα την έκθεσή μου, πνεύμα συνενετικό λοιπόν και σε μια συγκυρία ιδιαίτερη, ιδιάζουσα, μια συγκυρία που συζητήσαμε άλλωστε και χθε το απόγευμα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον πρόεδρο της Eurogroup. Και βλέπουμε ότι όλοι εδώ στην Επιτροπή μας ε, έχουμε δεσμευθεί να ε, συμβάλλουμε στο βαθμό που μπορούμε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τα ευρωπαϊκά όργανα στην αναζήτηση μέσων για αντιμετώπιση της κρίσης, να διαφυλάξουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, την βιωσιμότητα και αηφορία των δημοσιονομικών, των δημοσιονομικών, δηλαδή ανάκαμψη διαφύλαξη του κοινωνικού μοντέλου και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών που θα πρέπει να αποτελούν τους γνώμονες που θα μας καθοδηγήσουν στις συζητήσει μας. Δεν θα επισέλθω τώρα στις λεπτομέρειες. Την Τετάρτη έχουμε να δούμε τους σκιώδεις συγκητές και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να σα αναφέρω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συνένεση, είναι δυνατόν να βρούμε συνενετικές λύσεις γύρω από τα εξή στοιχεία. Οι τροπολογίε, από ό,τι φαίνεται τίνουν στις, ε, στο να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει να είναι αντικυκλικές οι ε, δημοσιονομικές παρεμβάσεις, δηλαδή τη στιγμή που θα υπάρχει έλλειμμα θα πρέπει να είναι σε θέση ε, ο δημόσιο προπολογισμό να... Ε, ρευστοποιεί το πλεόνασμά του, το, δημοσιονομικό του πλεόνασμα. Αντικυκλική όμως οικονομία σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν έχει ανακάμψει οικονομία. Θα πρέπει το κάθε κράτος μέλος και με βάση τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά να έχει στη θεσή του τα απαραίτητα περιθώρια χειρισμών έτσι ώστε να αναπτύξει τα απαραίτητα μέτρα στήριξης. Αντικυκλική πολιτική δηλαδή σημαίνει δύο πτυχές μία πτυχή σε περίπτωση ισορροπίας πλήρους απασχόλησης όπου βρίσκεται σε ανάκαμψη η οικονομία και μία πτυχή με στόχο την ανάκαμψη όπου θα αναφέρεται σε περίοδο κατά την οποία δεν αξιοποιούνται πλήρως ε, δεν χρησιμοποιείται πλήρω όλο το δυναμικό της παραγωγικότητας. Άρα λοιπόν εδώ βλέπω κάποιες προτάσεις για δημοσιονομικές δαπάνες ε, σε ορισμένες τροπολογίες. Δηλαδή όταν σε περίπτωση υποαπασχόλησης και ε, υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού θα πρέπει να σπρώξουμε την οικονομία σε μια ανάκαμψη. Βεβαίως χρειάζονται τα σχετικά μέτρα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, αλυσιτελούς δαπάνης, του αντίον μάλλον, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε στο δυνατόν πιο αποτελεσματικές δαπάνες και βλέπω ότι δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές όλες οι δημόσιες δαπάνες που ε, διατέθηκαν στην αντιμετώπιση κρίση. Και άρα θα πρέπει να γίνουν σχετικές μελέτες αποτελέσματος. Μια άλλη εστία συνένεσης που διαβλέπω εγώ αφορά τον ορισμό του τι θα πρέπει να είναι μια ανατασσόμενη οικονομία. Οι οικονομολόγοι λένε ότι η ανατασσόμενη είναι η οικονομία όπου η παραγωγή πρέπει να αξιοποιείται πλήρως. Το οποίο σημαίνει πως αξιοποιείται στην πραγματικότητα κατά 85% το παραγωγικά δυναμικό. Τώρα είμαστε κάπου στο 70 με 72% παρά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης και πέραν της ε, διελκυστήντας ως προς τα στατιστικά, ως προς το συγκεκριμένο ποσοστό δηλαδή της ανάκαμψης, θα μπορούσαμε πιστεύω να συμφωνήσουμε όλοι ότι όσο δεν αξιοποιούνται πλήρως οι παραγωγικοί πόροι, θα πρέπει να ενισχύουμε την πτυχή ανάκαμψη των αντικυκλικών οικονομικών πολιτικών. Και όταν πια αποδειχθεί ότι έχει ξεκινήσει πραγματικά η ανάκαμψη, τότε ασφαλώς θα πρέπει και να αξιοποιήσουμε και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού ή να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα όπως είπα νωρίτερα. Και ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ στην έκθεση αυτή είναι ότι βλέπω πιθανή μια συμφωνία, πιο δυσέβρατη ωστόσο, ε, στην συζήτηση για τα κριτήρια μου φαίνεται το απαραίτητο να βοηθήσουμε την Επιτροπή και να διακηρύξουμε ξεκάθαρα προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίες ε, κερδοσκοπούν αυτή τη στιγμή εις βάρος των εθνικών χρεών ότι μπορούμε να έχουμε ε, βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Στην οικονομική θεωρία όμως, όσο και αν ψάχνουμε, δεν βλέπουμε πουθενά κάποια συγκεκριμένη πρόταση από τους ειδικού ενός κριτήριου, κριτηρίου βιωσιμότητας των, ή ε, ανεκτού των, ε, του δημόσιου χρέους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσδιορίσουμε. Και εφόσον συμφωνούμε ως προς την ανάγκη για μια αντικυκλική πολιτική, η ιδέα είναι βεβαίως να ενισχύσουμε τα κριτήρια αυτά του Συμφώνου Σταθερότητας αλλά και άλλα κριτήρια, γι' αυτό είχα μιλήσει για μακροπρόθεσμα ε, ή βιώσιμες ε, οικονομικές, δημοσιονομικές πολιτικές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και να αντιμετωπιστεί το κριτήριο του ποσοστού διαρθρωτικού δανεισμού. Αυτές ήταν οι προτάσεις μου. Τις θεωρώ λογικές μέσα σε μια μακροοικονομική προσέγγιση. την οποία θα μπορούσα να χαρακτηρίσω μια συνθετική προσέγγιση. Και... βεβαίω βεβαίως υπάρχουν και άλλα σημεία από τις τροπολογίες, οι οποίες υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ενδεχομένως, αλλά πάντως στα τέσσερα πρώτα σημεία που σας ανέφερα πιστεύω ότι μπορεί να είναι επικοδομητική συζήτηση. Thank you. Uh, ευχαριστώ κύριος Χόκμαρκ. Thank you very much, uh, Madam Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή. Προσβλέπω να δω τη δουλειά που έχει γίνει με τις συμβιβαστικέ, αλλά θέλω να υπογραμμίσω πως πιστεύω πως οι συμβιβαστικέ λύσεις θα πρέπει να οικοδομηθούν επί τη βάση διαφόρων τροπολογιών που έχουν προέλθει από την ομάδα του ΕΛΚ και των φιλελευθέρων, γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, σε κάποια θέματα. Ελπίζω πως ο εισηγητής λοιπόν θα τα λάβει αυτά υπόψη για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από την Επιτροπή μας. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα κοιτάζουμε με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για την Ευρώπη ώστε να σταθεί στο στην εχμή των εξελίξεων για τις επόμενες δεκαετίες. Το είδαμε ότι το συζητήσαμε και πέρσι ότι το, στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε μια σαφή συνεπή στρατηγική αλλά και μια διασφάλιση ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια κρίση θα μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο τη δημόσια οικονομία μα. Και τα αποτέλεσματα εκείνη τη φορά ήταν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση με ακόμα πιο αυξημένε δαπάνε. Και για να είμαστε σοβαροί, ε, θα πρέπει να δούμε ότι αυτό δεν ήταν ε, ότι, το μέγεθος μάλλον της ανταπόκρισης γιατί στις χώρες που αυτή η επιλογή ακολουθήθηκε έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και είναι πρόβλημα γιατί θίγει την καρδιά του συστήματος πρόνοιας εκτός όλων των άλλων. Θα πρέπει να πω ότι όταν η Επιτροπή μας ε, συνάντησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό μπορούσαμε να δούμε ένα από τα αποτελέσματα ε, του ανεξέλεγκτου δημόσιου τομέα και του οικονομικού ε, της οικονομίας. Ε, τεράστια προβλήματα με τα ελλείμματα. Και δεν πρέπει εδώ να ξεγελαστούμε, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή κατά των δαπανών για την πρόνοια ή για τις νέες απασχόλησεις από την ε, δημόσια οικονομία που καθίσταται ανεξέλεγκτη, όπου δηλαδή αυξάνεται το έλλειμμα και το κρατικό χρέος επίσης αυξάνεται. Γιατί όταν αυξάνεται το κρατικό χρέος, το κόστος ε, εξυπηρέτησης των δοκίων ε, αυξάνεται αντίστοιχα και έτσι αποκλείονται άλλου είδους επενδύσεις. Γι' αυτό τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναπέσουμε στα ίδια προβλήματα και στα ίδιο λάθος. Και το τι κάνει ένα κράτος ως προς αυτή την ε, πτυχή επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους. Το βλέπουμε αυτό γιατί εντάξει συζητάμε τώρα την ελληνική οικονομία. Γιατί το κάνουμε, γιατί επηρεάζει την ανάκαμψη ολόκληρης της Ευρώπης. Και το ίδιο ισχύει και για διάφορα άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω πως είναι καλό που η συγκητής ε, μας δίνει εδώ μεγάλη ε, βιβλιογραφία, αλλά αν έχουμε δύο οικονομολόγους σε ένα, μια αίθουσα, θέλω να σας θυμίσω, προφανώ θα έχουμε και δύο διαφορετικές απόψεις και γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Με χαρά πάντα ακούω τις αναφορές στον κύριο Κέινς, αλλά νομίζω πως η γενική στάση είναι πως είναι πολύ εύκολο να αυξήσει κανείς τις δημόσιες δαπάνες και τα ελλείμματα και στον κόσμο του κυρίου Κέινς ήταν επίσης εύκολο να τα μειώσει. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο. Το είδαμε και στη δεκαετία του 70 και του 80 με τεράστια προβλήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία και μεγάλες επιπτώσεις στην απασχόληση. Προσβλέπω λοιπόν στην εξέβρεση διαφόρων συμβαστικών λύσεων, αλλά επίσης ότι αυτό θα γίνει επί τη βάση κριτηρίων που υπάρχουν ήδη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ορίσουμε νέα κριτήρια. Υπάρχουν τα κριτήρια του Συμφώνου σταθερότητα. Και έχουμε επίσης μα διδαχτεί από αυτή την κρίση ότι ένα από τα τεράστια σφάλματα που, που διαπράξαμε ήταν ότι δεν σεβαστήκαμε τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητα, γιατί αυτό οδήγησε στο γεγονός ότι αρκετά κρατημέλη που βρίσκονται στην αιχμή του κύκλου είχαν μεγάλα ελλείμματα, έχουν μεγάλα ελλείμματα και δεν μπορούν να ελέγξουν την οικονομία τους. Δεν μπόρεσαν μάλλον να ελέγξουν την οικονομία τους και να την συγκρατήσουν όταν ε, χτύπησε η κρίση. Αυτό που πρέπει τώρα να εξασφαλίσουμε είναι ότι δεν θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη με το κόστος τεράστιο για το χρέος ε, το οποίο στην ουσία ε, ε, καταργεί τις δυνατότητες για το κράτος προνοίας, τα διάφορα κοινωνικά πρότυπα που έχουμε στις χώρες μας, αλλά επίσης και ε, καταργεί τις δυνατότητες για επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις Πιστεύω πως αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να πω ότι όπως και η συγητής υποστηρίζει την δική του άποψη, φοβούμε ότι θα ανοίξουμε με αυτόν τον τρόπο ε, μια μεγάλη πόρτα για μια μεγάλη περίοδο, μακρά περίοδο μεγάλων ελλημάτων και ψηλών επιτοκίων. Το λέω αυτό ώστε να έχουμε ένα σημείο κίνησης. Έχω δει πολλούς φίλους από την ομάδα των φιλελευθέρων και των ε, ε, του ΕΛΚ και ευχαρίστω θα συζητήσω συμβαστικέ λύσει από αυτέ τι βάσει, αλλά θέλω να ζητήσω από τον εισηγητή να φροντίσει ώστε να έχουμε ε, μια σαφή εικόνα για την ανάγκη ελέγχου των δημοσίων οικονομικών της μείωσης των του δημοσίου χρέους, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για νέες επενδύσεις και κάλυψη του κόστους του κράτους πλονή. Θα πρέπει να διαβάσουμε βέβαια την βιβλιογραφία, αλλά να συζητήσουμε και τις διαφορετικές απόψεις που έχουμε. Είναι πολύ σημαντική πολιτική διαδικασία αυτή. Ε, um, Tack, värderade ordförande. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω σουηδικά, επιτρέψτε μου. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Είναι προφανές ότι ανησυχούμε και εμείς όπως και εκείνος όσον αφορά την εξέλιξη των δημοσίων δαπανών. Είναι επίσης προφανές ότι για πολλά πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά τους στόχους. Ο προλαλής εξάλλου αναφέρθηκε στην ε, φιλολογία που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα, στα θέματα που έχουν ε, γραφτεί από αυτού. Οι φιλελεύθεροι έχουν υποβάλει τροπολογίες. Και αυτό γιατί μας απασχολεί πολύ το θέμα της ε, ισορροπίας στις δημόσιες δαπάνες είναι προφανές ότι πρέπει να βγούμε από αυτήν την δημοσιονομική κρίση και ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δημόσιες δαπάνες ως έχουν σήμερα. Γεγονός όμως είναι ότι αν συνεχίσουμε προς τη σημερινή κατεύθυνση, τότε τα δημόσια χρέη κινδυνεύουν να φτάσουν σε ακραία ποσά. Κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει και την κοινωνία και τις ε, δαπάνες στους κοινωνικούς τομείς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί η έκθεση. Έκθεση που αποτελεί μια καλή βάση προς συζήτηση. Είναι καλό να έχουμε την προσέγγιση αυτή του εισηγητή. Έτσι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Όπως είπε όμως και ο Χάκμαν, υπάρχουν πολλές τροπολογίες από το ΕΛΚ και από τους φιλελεύθερους που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον εισηγητή. Για μένα είναι σημαντικό σε αυτή τη δουλειά να λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, δημογραφία στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση η γύρανση του πληθυσμού. Και αυτό πρέπει να το προσθέσουμε και στο γεγονός ότι η οικονομία μας βρίσκεται σε κρίση, σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και άρα χρειάζονται σοβαρά μέτρα. Για την Ελλάδα ισχύει αυτό που χρειάζονται θαραλέα μέτρα και πρέπει να αποφύγουμε άλλες χώρες να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθούν θαραλέα μέτρα παντού. Δεν πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του πιο αδύναμου, αντίθετα πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του περισσότερο ισχυρού, ώστε η ασθένεια να μην μεταδοθεί παντού στην Ευρώπη. Έρχομαι τώρα στα κριτήρια, στους δείκτες που μας επιτρέπουν να δούμε κατά πόσο μία οικονομία είναι σε ισορροπία, είναι βιώσιμη ή όχι. Ε, λοιπόν, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι βλέπουμε ξεκάθαρα πότε μια οικονομία δεν πάει καλά και πότε αντίθετα πάει καλά. Ξέρουμε ποιοι είναι οι δείκτες, υπάρχουν ήδη τα κριτήρια. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα σύμφωνο το οποίο ε, πέρασε από εξέταση, συμφωνήθηκε μεταξύ μας και πρέπει να τηρηθεί. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από την τήρηση του συμφώνου αυτού. Εν κατακλείδη, θέλω να αναφερθώ στη στρατηγική 2020. Είναι προφανές ότι η στρατηγική αυτή 2020 είναι ένα καλό μέσο που μας επιτρέπει να δώσουμε νέα όθηση στην οικονομία, για να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. Συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να τολμήσουμε να πάρουμε. Πρέπει να τολμήσουμε να στραφούμε προς θαραλές στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Και όπως έλεγε και ο Χάρκμαν πριν από λίγο, έχουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Θέλω να έχουμε επικοδομητική συζήτηση με τον εισηγητή από αύριο και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε καλές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε έκθεση που θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτή την τόσο ευαίσθητη κατάσταση στην οποία σήμερα βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σβέν και τώρα. Δεν καταθέσαμε τροπολογίες. διότι όλες οι διαδικασίες μας έφυγαν έξω από το πρόγραμμα. Θα ήθελα απλώς να κάνω μια παρατήρηση. Ότι είναι το ζήτημα αυτό το δημοσιονομικό, των δημοσιονομικών πολιτικών, πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε αφενός ε, τους μεν που λένε ότι, δεν υπάρχουν, ε, ότι το πρόβλημα είναι ότι παρεμβαίνουμε πολύ, ενώ από την άλλη ο εισηγητής λέει ναι παραπονιέστε αλλά δεν δίνεται και ορθολογικά κριτήρια. Και μάλιστα ε, ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Ίσως είναι δύσκολο να ανεβρεθεί κάτι τέτοιο στην ε, ε, μακροοικονομική θεωρία, αλλά αυτό το οποίο έχει ε, επηρεάσει τέτοια τη δική μας Επιτροπή ήταν η θεωρία η σχετική με την λογιστική. των δημόσιων των δημόσιων κονδυλίων, των δημοσιονομικών, δηλαδή όχι μόνο το τι υπάρχει στη θέση του κράτους, αλλά και το τι κάνουμε τα χρήματα αυτά, τα επενδύουμε, τα δαπανούμε μόνο. Εκεί είναι το κρίσιμο, πιστεύω, στοιχείο και επιχείρημα των συναδέλφων. Τι κάνουμε τα χρήματα αυτά. Αν υπάρχει λοιπόν μεγάλο ποσοστό πληθωρισμού και σημαντικό έλλειμμα, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δυστυχώ έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια νομίζω. Υψηλό χρέος και υψηλό έλλειμμα μαζί. Και στην τροπολογία 67, αν τη διαβάσουμε στην ε, γερμανική της έκδοση, δική σας νομίζω είναι, είναι κάπως ε, αστεία θα έλεγα. Εκεί που λέει δηλαδή ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικές, λύσεις, ε, εναλλακτικές και λύσεις για να ε, βελτιώσουμε τα ποσά της γενετικότητας. Νομίζω ότι είναι προφανής η λύση, αλλά δεν ξέρω, η διατύπωση κάπως μου φαίνεται αστεία εδώ πέρα θα πρέπει να την ε, κάνουμε πιο διακριτική. Okay, uh, Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Εσάια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να συμφωνήσω με τον κύριο Χάκλουντ και τον κύριο Χόκμαρκ. τους συναδέλφους από τις Σκανδιναβικέ χώρες του Δανών και του Σουηδό. στα όσα είπανε για, τις, ε, για τα δημοσιονομικά ε, των κρατών μελών και το δημόσιο έλλειμμα. Οι δημογραφικές εξελίξεις, οι δημογραφικές στατιστικές, η γύρενση του πληθυσμού φαίνεται να έχουν σημαντική επιρροή στην οικονομική κρίση. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται σε επίπεδο Φιλανδικού Υπουργείου ε, μια σειρά προτάσεων ε, για την αντιμετώπιση του ελλείμματος της Φινλανδίας που είναι 5,5% όπως παραδείγμα τη βελτίωση του επίπεδου των ε, δημοσίων υπηρεσιών. Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν η παράταση κατά τρία χρόνια του ορίου συνταξιοδότησης, όχι κατά δύο, κατά τρία. Επιπλέον, εφόσον αυξηθεί από 1,8 σε 2,3 παιδιά το ποστό γεννητικότητα των Φινλανδών γυναικών θα συμβάλλει επίσης η αύξηση αυτή ε, θετικά στην ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας μας. Μακροπρόθεσμα η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα παράδειγμα, ε, ακόμη ένα παράγοντα ανάπτυξης του ΑΕΠ. Πιστεύω σε εκ ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα στα, στις δημοσιονομικές επιλογές θα πρέπει να υπογραμμιστούν περισσότερο. Δεν αρκεί δηλαδή να λέμε ότι με την ανάληψη περισσότερου δανείων μπορούμε μακροπρόθεσμα να δώσουμε τις λύσεις στα δημοσιονομικά προβλήματα. Ευχαριστώ, υπερβάνος Περές. Ευχαριστώ πολύ. εφόσον από ό,τι φαίνεται είναι σε επεξεργασία αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες και υπάρχει γενικά καλή θέληση, θα περιοριστώ μόνο σε δύο ε, παρατηρήσεις. Η πρώτη που έχει να κάνει με την ε, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών ε, πολιτικών. Ε, νομίζω ότι εμείς ως Ευρωπαίοι καλούμεθα να διδαχθούμε και από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Η κρίση λοιπόν αυτή έχει οδηγήσει σε δηλώσεις και τοποθετήσεις και για το άσπρο και για το μαύρο. Καθένα λέει το ένα και μετά την άλλη μέρα λέει το αντίθετο. Και από την Ευρώπη και από την Αμερική ακούμε πολλέ προ αντιφατικέ θεωρίε. Πλην όμω, ε, το μαξιλαράκι πάνω στο οποίο μπορέσαμε να σταθούμε πέφτοντας και το, ήταν το γεγονός ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές ε, μέσα στην Ευρώπη τη στιγμή που οι ανταγωνιστές μας, Αμερικανοί και Κινέζοι, είχαν τελείως διαφορετική ε, συμπεριφορά ήταν αυτό που λέμε αυτόματοι σταθεροποιητές, τα συστήματα δηλαδή κοινωνικής προστασίας υγειονομικής περίθαλψης και ούτω, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι που μας κράτησαν δηλαδή από την κατάρρευση. Πλην όμω εδώ βλέπω στην έκθεση τον κίνδυνο να αποδυναμωθεί το δυναμικό αυτό χωρίς καν να προτείνεται μία λύση για αντικατάσταση με κάτι το πιο αποτελεσματικό ενδεχομένως. Και αυτό το βρίσκω επικίνδυνο γιατί δεν μπορούν να δημιουργηθούν θετικές δυναμικές, δεν αρκούν δηλαδή δημοσιονομικέ δημοσιονομικές πολιτικές για να εξασφαλίσουν για την Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της και τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και κάποια δείγματα που βλέπω από την Γενική ε, Διεύθυνση για την Απασχόληση νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν με σοβαρότητα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω κάθε πρόταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ε, ε, αποψήλωση του κοινωνικού μας μοντέλου, δηλαδή την κατάργηση των ε, αυτόματων αυτών σταθεροποιητών, θα ήταν για μένα πολύ επικίνδυνη. Και θα ήταν επικίνδυνη και ως προς την βιωσιμότητα των οικονομικών μακροπτών, μακροπρόθεσμα. Υπάρχει λοιπόν νομίζω ε, ανάγκη να συζητήσουμε ήρεμα, ψύχρεμα, γαλήνια, όλα αυτά τα πράγματα στην ώρα τους, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε και ποια είναι η εμπειρία που έχουμε εμείς από το παρελθόν. Το Σύμφωνο Σταθερότητα, σας ενθυμίζω, διορθώθηκε το 2005 με δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη είχε το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου και η δεύτερη την, ε, τον υπολογισμό με σημαντικότερο συντελεστή του χρέους από ότι το υπερβολικό έλλειμμα ή τουλάχιστον σε σχέση με το υπερβολικό έλλειμμα. Όλοι όμως το έχουν ξεχάσει τώρα. Τότε όλοι είχαμε χαρεί και νομίζω ότι ακόμη και ο Επίτροπος ε, ε, που το είχε αναλάβει το θέμα αυτό είχε, είχε συγχαρητηρίων, είχε θεωρηθεί πολύ σοβαρή η δουλειά του και η προσπάθειά του για την αναθεώρηση του συμφώνου. Πλην όμως τα προβλήματα που έχουμε τώρα κρίσιμο, ε, είναι σε κρίσιμο βαθμό προβλήματα που απορρέουν από αυτή την μεταρρύθμιση. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τα πράγματα στο κατά πρόσωπο και τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να τηρήσουν τις κύριες αρμοδιότητες προς την οικονομική τους πολιτική δεν μπορούν να λησμονούν ε, ότι η καταστολή δεν φέρνει αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει η δυστημία, τα κράτη-μέλη δεν είναι διαθεθειμένα να ε, κινηθούν όταν τα πράγματα ε, βαίνουν ε, άσχημα δεν μπορεί κανείς να επέμβει να τα διορθώσει, να τα διορθώσει την πορεία τους και επίσης γιατί οι κυβερνήσεις δεν κινούνται πριν τις υποχρεώσουν οι αγορές. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν το λαμβάνουμε τόσο πολύ υπόψη εδώ στη ζώνη του ευρώ είναι ότι η βιαιότητα των αγορών αντιδρά με καθυστέρηση με χρονική απόκληση δηλαδή και αυτό με μεγάλη και ένοχη ε, αφέλεια παραμελήθηκε από την ε, αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Την επίδραση δηλαδή των ε, αγορών. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα διαφορετικά. Τι μέσα χρειαζόμαστε για να λειτουργήσει το σύστημα αποτελεσματικά. Και εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσω να αναπτύξω αυτό το διάλογο με όλους τους συναδέλφους και τους ενδιαφερομένους δεν ε, λέω ότι δεν είναι καλή μέθοδος ε, το σύμφωνο σταθερότητας, γιατί πρέπει να διατηρηθεί και η αηφορία των δημόσιων οικονομικών και πρέπει να είμαστε θέση να ελέγχουμε το, ε, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίρρηση δεν έχω. Αλλά να έχουμε μια συνεργατική στρατηγική, μια ευφυή στρατηγική, μια στρατηγική η οποία θα φέρνει κέρδος για τους ωφέλη δηλαδή για τους ε, πάντες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μια ξερή στεγνή πολιτική μόνο, μόνο με κατασταλτικά δηλαδή μέτρα, γιατί δεν βοηθάει η καταστολή ε, την οικονομία. Πρέπει κανείς να θέλει να έχει το ευρωπαϊκό προϊόν για να το ε, στηρίξει. το συγγνώμη που μιλώ με τόση έμφαση και για τόση ώρα, αλλά είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερω γιατί έχει να κάνει με την με την προσέγγιση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Και ήθελα να δώσω αυτόν τον τόνο στη συζήτησή μα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή. Θέλω να τον συγχαρώ γιατί με την έκθεση αυτή μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε συζητήσεις πολιτικής φύσεως. Ως Ευρωβουλευτής από το ΕΛΚ πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με την παρουσίαση του κύριου Χάτμαν και πρέπει να πω ότι τα σχόλιά μας πρέπει να είναι πολιτικά. Αν δούμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για παράδειγμα, η ανάλυση μας πρέπει να αφορά τα δύο σκέλη. Και την σταθερότητα, βεβαίως, αλλά δεν θα πρέπει από την άλλη να ξεχνάμε το άλλο σκέλος, που είναι η ανάπτυξη, που είναι επίσης αναγκαία για την οικονομία. Όσον αφορά λοιπόν την εφαρμογή του συμφώνου, ας πάρουμε για παράδειγμα τη δικιά μου χώρα, την Πορτογαλία. Εκεί για πολύ καιρό συζητήσαμε για το έλλειμμα και ξεχάσαμε το δημόσιο χρέος με αποτελέσματα πολύ σοβαρά. Όσον αφορά τα επιτόκια και την, ε, τους μελλοντικού φόρους, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να δούμε, γιατί κάποιος θα πρέπει να πληρώσει τελικά το λογαριασμό. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε τι γίνεται με το δημόσιο χρέος, αλλά πρέπει συγχρόνως να δούμε τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο και τι κάνουν τελικά τα κράτη-μέλη και τι δεν κάνουν. Πρέπει να σκεφτούμε την αποτελεσματικότητα. Τα ταμεία αυτά χρησιμοποιούνται, τα ευρωπαϊκά καλά. Πρέπει να καταλήξουμε σε πολιτικές επιλογές. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Μεγάλο, σοβαρό. Το ξέρουμε εξαιτία ε, της ε, δημογραφικής εξέλιξης στην Ευρώπη. Σήμερα στην Ευρώπη η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Θα έπρεπε να αλλάξει. Έχουμε λοιπόν υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Τέλος, ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την αντιμετώπιση των δημοσίων ε, δαπανών όταν αυτές είναι υπερβολικές. Πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα για όλες τις χώρες και πρέπει να αναλύσουμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τις στρατηγικές εξόδου από την κρίση, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να πάμε πιο μακριά από ό,τι μας επιτρέπουν οι σημερινοί κανόνες. Όσον αφορά τώρα τους δείκτες για μια οικονομία σε ανάκαμψη, εδώ τα κριτήρια πρέπει να είναι ελαστικά. Η κατάσταση είναι διαφορετική στις διάφορες χώρες. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε άκαμπτοι όταν μιλάμε για το τέλος της κρίσης. Συχνά ξεχνάμε μια πολιτική που είναι η φορολογική πολιτική. Πολλές φορές σκεφτόμαστε την ανταγωνιστικότητα, και έτσι βλέπουμε τη φορολογική πολιτική των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως την ανταγωνιστικότητα αυτή πρέπει να τη δούμε και σε σχέση με χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φροντίσουμε για μια πραγματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στο μέλλον πρέπει να φροντίσουμε για σταθερότητα και για ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε, ο κύριος ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με το κλίμα της ε, αντιμετώπισης αυτών των μακροοικονομικών πολιτικών. Έχω εν γέννη ε, την τιμή να είμαι μέλος εδώ της Επιτροπής μας από το 1999 μέχρι σήμερα και ασφαλώς αυτήν ε, μακροχρόνια σταδιοδρομία μου έχω δει ότι και εκείνοι που λένε ότι είναι καλύτερα και εκείνοι που είναι χειρότερα τα πράγματα έχουν δίκιο καθένας κάθε φορά και πιο πολύ φάνηκε ότι είχαν δίκιο τα τελευταία δέκα χρόνια ιδιαίτερως εκείνοι που έλεγαν ότι το κράτος ε, δεν πρέπει να παρεμβαίνει και ότι ε, το μερίδιο του κράτους ε, στην, ε, στο ΑΕΠ είναι πολύ υψηλό. Η Επιτροπή άλλαξε όμως ριζικά, όπως και οι πολιτικές δυνάμεις, εκεί όπου άρχισαν οι ίδιες αυτές πολιτικές δυνάμεις να κρατικοποιούν τράπεζες, επιβαρύνοντας έτσι τον φορολογούμενο, δηλαδή ο φορολογούμενος ήταν εκείνος ο οποίος ε, βρίσκεται διέξοδο, ε, πλήρωνε τα σπασμένα της κρίσης και ε, πλήρωνε αυτούς που έπαιζαν πόκερ με τα δημοσιονομικά του έτσι ώστε να βγουν από την κρίση. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Κράτη-μέλη τα οποία είναι υπερχρεωμένα και δεν ξέρουν πώς μπορούν να οργανώσουν την οικονομική τους πολιτική. Πρόκειται για μια εικόνα η οποία δεν ε, είναι τελείως λάθος. Οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση και να έχει κανείς, λίγο πολύ συνοψίζει την πραγματικότητα αυτή η εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν. Πάνω απ' όλα δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό το πράγμα δεν πρέπει να απαγορευθεί να διατυπώνουμε τις κρίσιμες ερωτήσεις. Ε, η οικονομική πολιτική δεν θα πρέπει να είναι απλώς μια βολική τοποθέτηση. Πρέπει να κοιτάμε τα δύσκολα θέματα. Και ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε συμβαστικές λύσεις ε, για να προωθήσουμε την έκθεση καλές συμβαστικές λύσεις, πρέπει να διατυπώσουμε τα κρίσιμα ερωτήματα, τα ενοχλητικά ακόμα ε, ερωτήματα, να προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από τα, από τα λάθη του παρελθόντος και να ε, αναθεωρήσουμε το ρόλο του κράτους, γιατί κανείς αυτή τη στιγμή δεν λέει ότι το κράτος ε, κάνει σημαντικές προσπάθειες για να εξηγιάνει την οικονομία του και να βγει από την κρίση. Ε, θα ήταν καλό να βρούμε μια καινοτόμο προσέγγιση μέσα από αυτή την ε, νέα έκθεση, μια νέα προσέγγιση που να προσφέρει και στην Επιτροπή μας μια φωνή, τη δυνατότητα δηλαδή να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ευχαριστώ Κλίντς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα μια παρατήρηση. Δεν είμαι σκιώδης ηγητής και δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό εντατικά, αλλά φυσικά πρόκειται για θέματα που μας καίνε όλους. Δημοσιονομικά, χρέη, υπερβολικά χρέη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν είναι ε, ασθενική η ανάπτυξή μας δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα ε, δημοσιονομικά μας, δεν μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε και βλέπουμε επίσης ότι ακόμη και αν φτάσουμε στο δυναμικό της ανάπτυξής μας πάντα μένει ανεπαρκές αυτό για να ε, εξηγιάνει τα δημοσιονομικά μας. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν αρκεί αυτό για να ε, φτάσει ο προπολογισμό σε, σε ένα ισοζύγιο τέτοιο που να είναι σύμφωνο με τα κριτήρια του Μάστριχτ. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με το δυναμικό της ανάπτυξης, αλλά έχουμε να κάνουμε και με, το, με πόσο σοβαρότητα ε, ρυθμίζουμε την ε, οικονομική μας ζωή και η δραστηριότητα. Και εγώ παραπέμποντας στην εμπειρία μου από τη Γερμανία, θα θέλω να πω ότι το 50% περίπου το διαθέτουμε μόνο για τον κοινωνικό τομέα και το τομέα της ε, απασχόλησης ε, το 50% του προϋπολογισμού μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό το σύστημα και θα πρέπει να το τροποποιήσουμε. Θα πρέπει να το σχεδιάσουμε διαφορετικά. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση ένα έλλειμμα να το εξετάσουμε κατά κάποιο τρόπο σαν ε, τις επενδύσεις στο μέλλον. Δηλαδή, οι επενδύσεις που θα κάνουμε να είναι αυτές τις οποίες θα χρειαζόμαστε και στο μέλλον και θα μας οδηγήσουν προς μια ανάπτυξη. Εάν όμως κάνουμε ε, δαπάνες, χρεωνόμαστε κατά τρόπον ώστε να μην έχουμε ε, επένδυση ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό το οποίο δαπανούμε να μην αποτελεί επένδυση για το μέλλον, τότε προφανώς μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα νερά και βαθιά κρίση. Ευχαριστώ κύριο Σικλούνα. Και αν ε, τυχόν ε, έχει κανείς παρατηρήσει τη διαφορά, ε, το ένα ρολόι πάει πίσω πέντε λεπτά, ενώ το άλλο πάει πίσω τέσσερα λεπτά, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περισσότεροι εξημών. Είμαστε νομοταγείς πολίτε. Όχι επειδή υπάρχει αστυνομία και κάθε πρωί βλέπουμε το ίντερνετ και ε, βλέπουμε τι λένε οι δικηγόροι και οι νομικοί και φοβόμαστε. Το κάνουμε επειδή είναι κοινή λογική. Παρομοίω λοιπόν θα ήθελα να τονίσω το θέμα τη ε, καλή πρακτική και τη καλή διαχείριση. Η βιωσιμότητα τη δημόσια οικονομία ε, είναι αντίστοιχη με την βιωσιμότητα των συστατικών της. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε καλή φορολογία, είτε έμεση είτε άμεση. Υπάρχουν πολύ καλές πρακτικές ε, σε αυτό το τομέα. Το ίδιο όσον αφορά τη βιωσιμότητα της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων. Και μετά, πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν και τα θεσμικά ζητήματα όπως η διαφάνεια, η απόδοση λογαριασμών και η καλή πρακτική. Δεν νομίζω λοιπόν πως οποιοδήποτε κανόνας μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Αυτά βρίσκονται, οι κανόνες υπάρχουν για τους ε, εκτός ε, συναγωνισμού, για τους παραβάτες κτλ. Αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη, ε, ιδιαίτερα σε δημοκρατικές χώρες υπάρχει πάντοτε η πίεση να δαπανά κανείς περισσότερα και να φορολογεί λιγότερο. Όμω, τα περισσότερα θέλουν να δουν ποια είναι η καλύτερη πρακτική και τι κάνουν οι, τα αντίστοιχα κράτη και οι εταίροι του. Και δεν πρέπει να το παραμελούμε αυτό το ζήτημα. Είναι βέβαια, επισχύει βέβαια ο ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, αλλά δεν είναι και τόσο τη μόδα λόγω τη κρίση και των προβλημάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ωστόσο, δεν νομίζω πως θα πρέπει να την αγνοήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο τελευταίος ομιλητής μας, οπότε επανέρχομαι στον εισηγητή. Έχετε τέσσερα λεπτά πριν φτάσουμε πραγματικά στις, 4, στις ε, μισή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να καθησυχάσω το σκιώδη συγητή από το ΕΛΚ όσον αφορά την εισαγωγή μου. Ήθελα ακριβώ να ξεκινήσω από τις τροπολογίες σας και τα δύο πρώτα σημεία τα οποία εξέθεσα είχαν απορρέουν ακριβώς από την μελέτη των δικών σας προτάσεων. Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για την αναγκαιότητα πολιτικών αντικυκλικών και εγώ δεν αναφέρομαι στον Κέινς. Σε αυτά που εσείς γράφετε, που λένε ότι όντως πρέπει να δούμε τα πλεονάσματα και την χρέωση. Αλλά συμμετρικά, γιατί βλέπετε ότι στο κάτω σημείο του κύκλου, όταν η οικονομία δηλαδή γυρνάει με πολύ χαμηλή απόδοση, πρέπει να κάνουμε αυτό που ονόμασε η ε, κυρία Μπερές ε, αυτόματους δείκτες. Οπότε, αυτόματους μάλλον σταθεροποιητές. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Το δεύτερο σημείο τώρα για το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι η αξιολόγηση της φορολογικής δαπάνης. Επ' αυτού πολλοί και από τη δεξιά και από την αριστερά και από το κέντρο επέστησαν την προσοχή μας στην αναγκαιότητα να μην σπαταλάμε το δημόσιο χρήμα. Και όλα τα περί φορολογικών δαπανών νομίζω ότι μπορούν να μας βρουν σύμφωνος. Τώρα, συμφωνία για τα κριτήρια, τέλος. Εγώ δεν ήρθα στο κοινοβούλιο για να κάνω θεωρία, αλλά για να κάνω πολιτική. Γι' αυτό είμαι εδώ. Η συζήτηση λοιπόν που έχουμε για τα κριτήρια δεν είναι μόνο θεωρητική συζήτηση, είναι κύρια πολιτική συζήτηση. Όταν τονίζω λοιπόν την ανάγκη να συμπληρώσουμε τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας, δεν αμφισβητώ το Σύμφωνο Σταθερότητας, όχι. Είμαι στην ίδια γραμμή από την αρχή. Σέβομαι το Σύμφωνο Σταθερότητας όσον αφορά την αναθεωρημένη του εκδοχή του 2005. Δεν είμαι από αυτούς που αμφισβητούν την αναθεώρηση αυτή του 2005 του Συμφώνου Σταθερότητας. Όχι. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όταν όμως λέω ότι πρέπει να συμπληρώσουμε τα σημερινά κριτήρια, τα οποία είναι ασαφή μερικές φορές, στην δεκαετία του 80 που είχαμε το μισό έλλειμμα και χρέος από τις διάφορες χώρες. Άρα λοιπόν το πλαίσιο εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικό. Και η λιτότητα που χρειαζόταν τότε ήταν διαφορετική. Άρα λοιπόν εγώ δεν είμαι υπέρ της καταστολής όπως κάποιοι λέγανε νωρίτερα. Όντως δεν λειτουργεί, δεν κάνει καλό, κανείς δεν καταφέρει να τηρήσει το σύμφωνο σταθερότητα στη σήμερα ημέρα. Το πραγματικό πρόβλημα σήμερα είναι τι μήνυμα στέλνουμε εμείς στις δημοσιονομικές αγορές σε ένα πλαίσιο όπου όλοι αναγνωρίζουν ότι οι οικονομικές αγορές δεν εκτίμησαν καλά τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με το ενεργητικό κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει και υπερεκτίμηση του χρέους. Αν βάλουμε απ' έξω την Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρος ότι η Ισπανία έκανε ό,τι καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Οι αγορές βάλουν και την Ισπανία σήμερα. Λοιπόν, τι μήνυμα εμείς στέλνουμε στις αγορές, τι μήνυμα στέλνουμε στους ε, οργανισμούς αξιολόγησης. Δεν έχω απάντηση, αλλά λέω να το σκεφτείτε. Τι μήνυμα μπορούμε να στείλουμε στις οικονομικές αγορές για να τους δείξουμε ότι αντίθετα με αυτό που νομίζουν η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών δεν είναι τόσο καταστροφική. Είμαστε στο κάτω σημείο του κύκλου, εγώ αυτή την αίσθηση έχω γιατί στο 70% χρησιμοποιούμε τις δυνατότητε παραγωγής, υπάρχει πρόβλημα ε, μη επαρκούς ζήτηση στην Ευρώπη. Αλλά αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε νομίζω πιο καρποφόρα την Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πάντως για τις επικοδομητικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των τροπολογιών είναι ότι περιμένουμε 27 ε, Απριλίου για να μπορέσουμε να την στείλουμε στην Ολομέλεια τον Μάιο, στη δεύτερη Ολομέλεια και να είναι έτοιμη για το Συμβούλιο του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ. Και προχωράμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης και θα βγω λίγο για να βρω τον κύριο Κωνστάνσιο. Μισό λεπτό λοιπόν υπομονή. you very um, ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε τώρα σε μια ανταλλαγή απόψεων με τον υποψήφιο για την Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Βίτορ Κωνστάνσιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για 15 λεπτά και έπειτα θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσει ε, θα είναι όπως γίνονται για τον νομισματικό διάλογο. Ήδη έχετε δηλαδή τον κατάλογο με την ε, σειρά με την οποία θα υποβάλλετε τις ερωτήσεις σα. Δίνω λοιπόν το λόγο αμέσως στον κύριο Κωνστάσιο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα και πάλι ενώπιον της Επιτροπής σας για αυτή την ακρόαση που αποτελεί τμήμα της διαδικασίας ε, του διορισμού μου στην Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, στην πρόσφατη μου παρουσία ενώπιον της Επιτροπής σας για μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων είχα την ευκαιρία να συνοψίσω στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις ε, την θέση μου για κάποια από τα πιο σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την νομισματική πολιτική. Έπειτα εξέφρασα τις απόψεις μου για την φύση της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον νόημα του δευτερεύοντος στόχου, όπως ορίζεται στη συνθήκη, τα βασικά στοιχεία της ε, νομισματικής μας στρατηγικής, το ρόλο της ε, νομισματικής σταθερότητα και των τιμών των ακινήτων στην νομισματική πολιτική και τέλος ε, συζήτησα την αξιολόγησή μου των πληθωριστικών κινδύνων στην παρούσα κατάσταση. Σκοπός μου δεν είναι να καλύψω αυτά τα θέματα στη σημερινή μου δήλωση, αλλά εν ώψη σημασία θα ήθελα να προτείνω το γραπτό μου εισηγητικό κείμενο στην προηγούμενη επόμενη μας ε, συνάντηση θα μπορούσε να προσαρτηστεί σημερινές, ε, στα σημερινά σας πρακτικά. Σήμερα θα εστιάσω την προσοχή στα αρχικά μου σχόλια στα θέματα ρύθμιση και δημοσιονομική σταθερότητα. Όπω ανέφερε και την περασμένη φορά, η ανάγκη να αποφευθεί η ρήξη στη λειτουργία του δημοσιονομικού συστήματο ε, έχει να κάνει και με την νομισματική πολιτική. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί από τι κεντρικέ τράπεζε, γιατί τα χρηματοπιστωτικά ε, θεσμικά όργανα, οι θεσμοί μάλλον, είναι πολύ σημαντικοί για την οικονομία και για την διαβίβαση ε, τη ίδια τη νομισματική πολιτική ότι η κρίση είναι ένα παράδειγμα μαζικών αναταράξεων στον δημοσιονομικό τομέα. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά διδάγματα που θα πρέπει να αποκομίσουμε από αυτή την κρίση. Πρώτον, ο δημοσιονομικό τομέας δεν είναι δεν αυτοισορροπείται ούτε αυτοδιορθώνεται. Ένα τέτοιο ε, χρηματοπιστωτικό τομέα μπορεί να δημιουργήσει κρίση ε, ο ίδιο, αυτογενή. Ε, οι εκτεταμένες περίοδοι μεγάλης ανάπτυξης ε, στην ε, πίστη και στην χρέωση οδηγούν σε άνθηση των τιμών των ακινήτων που και πάντοτε καταλήγουν σε κρίση. Και τέλος, ο χαμηλός πληθωρισμός στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών δεν αρκεί για να εγγυηθεί την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτά τα μαθήματα τα έχουμε μάθει και τα έχουμε ξεχάσει αρκετές φορές ε, κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας. Ε, η κακή συμπεριφορά των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η απορρίθμιση και διάφορα σκοτεινά κίνητρα δημιούργησαν μια τέτοια καταιγίδα που για πολύ καιρό θα συνεχίζει να προκαλεί ανεργία και χαμηλή ε, μεγέθυνση. Άρα λοιπόν το θέμα είναι το εξή. Μπορούμε εμεί να εφεύρουμε τέτοια μέσα και θεσμού ώστε να μπορέσουμε να αντιθασέψουμε αυτέ τι ε, ακρότητε τη οικονομία χωρί να θέτουμε σε κίνδυνο τον ρόλο τη. Μια αισιόδοξη άποψη ε, είναι ότι μπορούμε να βασιστούμε σε μια θετική αξιολόγηση της κρίσης και όλα αυτά έχουν ε, γεμίσει τα γραφεία μας. Θα ήθελα να σας αναφέρω διάφορες τέτοιες προτάσεις με διάφορες σύντομα σχόλια, γιατί πολλά από αυτά είναι ήδη ε, γνωστά τη πάση. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι τα δικά μου βασικά σχόλια και αργότερα θα αναπτύξω περισσότερο ορισμένες προτάσεις που πιστεύω πως δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη, δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί. Πρώτον, η δημιουργία μιας μακροπροληπτικής ευθύνη που θα ανατεθεί σε ένα υπάρχον ή ε, νεοτεχθέν ε, ίδρυμα ή οργανισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή που προκύπτει ε, μια κρίση από την, που, που οφείλεται στη γενική κατάσταση της οικονομίας ή των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς αρμοδιότητες θα δώσουμε σε ένα τέτοιο θεσμό. Δεύτερον, η εισαγωγή νέων προδιαγραφών με περισσότερο και καλύτερο κεφάλαιο με βάση τις προτάσεις της ε, Επιτροπής της Βασιλείας. Ε, τρίτον, η μείωση των... Ε, της υπερκυκλικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου μέσω ενός συστήματος ε, ε, κεφαλαικών φραγμών ή δυναμικών προβλέψεων ή αποθεμάτων. Στην πρώτη μέθοδο απαιτείται κεφάλαιο το οποίο θα αυξηθεί στα καλά χρόνια ενώ θα μειώνεται στις άσχημες χρονιές. Εγώ προσωπικά προτιμώ τις δυναμικές προβλέψεις αλλά Οποιοδήποτε από αυτές τις μεθόδους είναι προτιμότερη από τη σημερινή κατάσταση. Η διόρθωση τώρα των ε, λογιστικών ε, προδιαγραφών που αυτή τη στιγμή ε, επιτρέπουν κέρδη χωρίς πραγματικά κεφαλαιακά κέρδη σε περιόδους άνθησης ε, και υπερβολικές, ε, ε, υπερβολική μείωση στα κέρδη στις κακές χρονιές. Πάλι λόγω των μη πραγματικών κεφαλαϊκών απολειών ή ζημιών. Χρειάζεται λοιπόν η ανάγκη για ένα αποθεματικό με βάση τον οικονομικό κύκλο όπως προτείνεται στην έκθεση Turner, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να υπολογιστούν με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και προηγουμένως στο τρίτο σημείο που σας ανέφερα, γιατί είναι απαραίτητο να επηρεάζονται οι λογιστικές εκθέσεις ώστε να αποφεύγονται οι πτυτικές, τα πτυτικά κέρδη που επηρεάζουν τις ε, τιμές των μετοχών αλλά και τα κέρδη των χρηματοπιστωτικών θεσμών. Έπειτα, η εισαγωγή ενός ανώτατου απόλυτου ποσοστού μόχλευσης, η εισαγωγή νέων ποσοστών ρευστότητας όπως προτείνει η Επιτροπή της Βασιλείας, επαγόρευση απαγόρευση σκιώδους τραπεζικού τομέα και η ενθάρρυνση και η ενίσχυση μάλλον των ε, παγιωμένων λογιστικών κανόνων. Ε, στη συνέχεια αυστηρότεροι ε, κανόνες όσον αφορά την τιτλοποίηση. Τα όσα συνέβησαν με τα ανυπόθηκα ομόλογα, της ασφαλίσεις έναντι της αθέτησης πληρωμών, το CDO ήταν πραγματικά τρομακτικό και δεν πρέπει να ξανασυμβεί ένα-ένα ε, το σημείο είναι ο περιορισμός της εμπιστοσύνης στις, ε, στους οργανισμούς αξιολόγησης που συνέβαλαν στην υπερκυκλικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και έπαιξαν πολύ αρνητικό ρόλο στην ε, κρίση των ενυποθήκων δανείων. Η απλή καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του μπορεί να μην αρκεί για να διορθωθεί η αποδοτικότητά τους και η απόδοσή τους η εισαγωγή νέων κανόνων ε, ώστε να διορθωθούν και να μπορούν να, να μάλλον ε, τα σκοτεινά αυτά κίνητρα που, που αναφέραμε με τις ε, υπερβολικές βράχοι πρόθεσμες προπτικές. Γενικά όλα αυτά έχουν ε, συμπεριληφθεί στο, στις προτάσεις και τις δευτήριες γραμμές ε, του Συμβουλίου Οικονομικής Σταθερότητας και εκρίθηκαν από τους, ε, την ομάδα των 20, του G20. Ωστόσο θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά τέσσερις πτυχές που θεωρώ πιο σημαντικές ή που δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς. Το πρώτο σημείο αφορά την αξιολόγηση του κατά πόσο οι νέοι κανόνες επαρκούν ώστε να παρεμποδίσουν τις, τις υπερβολές της ε, χρηματοπιστωτικής αγοράς και κατά πόσο η μακροπροληπτική διαδικασία εφαρμόζεται με αυτό το στόχο. Η απάντησή μου την είναι ναι, θετική, γιατί μέσα όπως ε, η χρήση του δεύτερου πυλώνα ε, οι, άλλες, ε, οι άλλα μέσα μπορούν να αρκέσουν για ένα τέτοιο έργο. Τώρα, όσον αφορά την μακροπροληπτική πολιτική, φαίνεται λες και σε όλες τις χώρες ε, το θεσμός που θα αναλάβει κάτι τέτοιο θα περιορίζεται στο να εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις. Στην Ευρώπη η πρόταση συστάση του ESRB, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου με τη συμπερίληψη της Κομισιόν και των ε, τριών εκπροσώπων ε, των κεντρικών τραπεζών μπορεί να διασφαλίσει την εγγύηση, του, να διασφαλίσει τον συντονισμό ανάμεσα στα επίπεδα μικρο και μάκρο Ελπίζουμε πως έτσι η μακροπροληπτική λειτουργία δεν θα περιοριστεί μόνο σε κηρύγματα προειδοποίησης ε, και χτύψεις. Εγώ παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτησή σας ε, στην Επιτροπή σα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κίνδυνο Κινδύνου και πιστεύω πω πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα για την αποτελεσματική λειτουργία αυτού του νέου οργάνου. Καταρχήν, η Διοικητική Επιτροπή του θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύσταση του Γενικού Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να αποφεύγονται οι εντάσει. δεύτερο αφορά στην ανάγκη να διατηρηθεί η προτινόμενη σύσταση του Συμβουλευτική τεχνική επιτροπή, γιατί βασικό της ρόλο είναι να προετοιμάσει τις εργασίες του Γενικού του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι πιο αποτελεσματική να αποτελείται από ανθρώπους που εργάζονται μέσα στα θεσμικά όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για το, τη ρύθμιση και την εποπτεία ε, Μπορεί αυτό να προσθεθεί απλώς στην ε, ε, αρχιτεκτονική χωρίς να εξαλειφθεί το συστατικό της προπαρασκευαστικής εργασίας για το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δεύτερο παρατήρηση που θέλω να κάνω σχετίζεται με την ανάγκη να μεταφερθούν ε, όλα αυτά τα παράγωγα, τα πιστοτικά παράγραφα, ιδιαίτερα το εμπόριο στα CDS που είναι οι ασφαλίσεις για θέτηση πληρωμών ε, και τα πριμ που τόσο ευρέως χρησιμοποιούνται, αυτά είναι κάπως ακατανόητα προϊόντα και συνήθως ε, οι συναλλαγές γίνονται κάτω από το τραπέζι. Ε, είναι απλά αναφορές που στέλνονται σε μια ιδιωτική εταιρεία που ξεκίνησε να φτιάχνει στατιστικές το 2001. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς λειτουργεί το πράγμα και οι παίκτες δεν είναι γνωστοί. Και επειδή απλώ είναι αναφορές, είναι, είναι δηλαδή τιμές σε μια ανοργάνωτη αγορά, οι θεσμοί, θεσμοί που κάνουν τέτοιου ε, ε, δίνουν τέτοιου είδου, μάλλον τιμές, δεν είναι υποχρεωμένε να τα δηλώνουν όλα αυτά. Ο Μάιλον σόλ, που είναι ένα είδος ε, νονού για τα παράγωγα προϊόντα, είπε πέρσι. Η λύση είναι να εκραγεί ή να καεί η αγορά αυτών των παραγόγων, τα CDS και τα swap και τα διάφορα δεδομένα προϊόντα και να ξεκινήσουμε αυτού και από την αρχή. Θα πρέπει επίσης σοβαρά να σκεφτούμε τη δυνατότητα της απαγόρευσης της πώληση αυτών των μέσων που επιτρέπει μόνο στα θεσμικά όργανα της αγοράς να κάνουν τέτοιου είδους ε, συναλλαγές ως δραστηριότητα τύπου hedge fund. Η τρίτη πτυχή που θέλω να αντιμετωπίσω είναι εκείνη η κολοσσή που θεωρείται ότι δεν μπορεί να χρεοκοπήσουν ε, η ύπαρξη τέτοιου είδους κολοσσών ε, που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταρρεύσουν, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα ηθικού τύπου που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη συμπεριφορά. Και δεν υπάρχει συμφωνία διεθνώς για το πώς να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ε, ε, τεράστιοι οργανισμοί. Αυτό ίσως ακόμη περισσότερο να είναι προβληματικό μετά την κρίση. Δεν έχω τη λύση, αλλά δεν πιστεύω πως μπορεί να λυθεί μέσω μιας πολιτικής συστηματικού κατακαιρματισμού μεγάλων ε, τέτοιων εταιριών ή κολοσσών και με τη λύση της προστασίας μόνο των μικρών ε, τραπεζών και τη διάκριση μεταξύ των ε, επενδυτικών τραπεζών και των υπολείπων. Υπάρχει λοιπόν ένας κατάλογος προτάσεων ε, που έχουν γίνει, ορισμένες από αυτές ε, ε, εξετάζονται και μέσα στο πλαίσιο προετοιμασίας σχετικής νομοθεσίας δεν θα σας παραθέσω όλο τον κατάλογο. Αλλά πιστεύω ότι η χρήση αυτών των μέσων που δεν αποκλείουν το ένα το άλλο είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ε, δηλαδή απαιτήσει για τα κεφάλαια, οι ασφαλίσεις φυσικά και ιδίως η δημιουργία ενός ειδικού ε, καθεστώτος ε, επίλυσης ε, των ε, προβλημάτων ή ε, εκαθάρισης καλύτερα θα το λέγαμε, δηλαδή για εκείνα τις, επιχειρή... τις ε, τράπεζες ή τους θεσμούς που δεν μπορούν, οργανισμούς που δεν μπορούν πλέον να σταθούν και πρέπει να διαλυθούν, όπως έγινε ας πούμε τη General, General Motors. Το υπεύθυνο θεσμικό όργανο, για, θεσμός, οργανισμός για τέτοιο είδος ε, ρόλο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε έναν ταμείο αναδιάρθρωσης ή εκαθάρισης. Το τελευταίο πρόβλημα που δεν έχει ακόμα επιληθεί αφορά την επίλυση κρίσης ή <clears throat> όσον αφορά τους διεθνείς οργανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βρεθούν συντονισμένες λύσεις σε αυτό. Το βασικό εμπόδιο αφορά την μοιρασιά του κόστους όσον αφορά την επίλυση της κρίσης. Όπως έγραψα στις απαντήσεις μου προς το ερωτηματολόγιο σας, πιστεύω πως εν τέλει μια πραγματικά ευρωπαϊκή λύση θα απαιτήσει και ένα ευρωπαϊκό ταμείο ε, εγκαθάρισης ή επίλυσης των κρίσεων, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξει λύση. Μάλιστα την, τελευταία, την περασμένη Παρασκευή διαπίστωσα πως και ο Επίτροπος Μπαρνιέ κατευθύνεται προς την ίδια... Ε, έχει μάλλον τον ίδιο προσανατολισμό. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω πως χρειάζεται ε, περισσότερη εναρμόνιση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα αφαιρεγγιότητας. Τέλος, να σας πω κάτι σχετικά με τον αντίκτυπο όλων αυτών των προτινόμενων μέτρων. Μπορεί, κάποιοι λένε ότι η υπερβολικά μεγάλη νομοθεσία, πολλή νομοθεσία μπορεί να σκοτώσει τελείως την οικονομία. Όμως, ε, πιστεύω πως δεν θα υπερέβαλε κανείς ε, λόγω της κρίσης που διανύουμε να γίνουν τέτοιες ε, ρυθμιστικές προσπάθειες. Ε, ωστόσο θα πρέπει να απευθυνθεί ο κίνδυνος όσον αφορά τον χρονισμό της εφαρμογής τους. Η ταχεία εφαρμογή όλων των μέτρων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τις απαιτήσει περί κεφαλαίων, μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς που να, να καθυστερήσουν την οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει ωστόσο να είναι αποφασιστική η δράση και η νομοθεσία όσον αφορά το περιχώριο περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων, όσο θα πρέπει να είναι και συνετή ε, η στιγμή της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις ερωτήσεις σε ένα λεπτό, αλλά θα ήθελα πριν από αυτό να σας ανακοινώσω ότι οι βοηθοί θα πρέπει να κάθονται στις θέσεις όπου είναι σημειωμένες για τους βοηθούς. Δεν θα πρέπει να κάθονται στις θέσεις στα έδρανα των των βουλευτών και κυρίως όχι δίπλα τους και να συζητούν μαζί τους κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Χάνς Πίτερ Μάρτιν και η κυρία Ντάτη, παρακαλώ, ε, έχετε τους βοηθούς σας δίπλα σας, ε, παρακαλώ να μετακινηθείτε. Ναι, ούτε καν βάλετε τα ακουστικά σας, δεν μπήκατε καν στον κόπο να βάλετε τα ακουστικά σας για να μ' ακούσετε τι σας λέω. Θα συνεχίσουμε όταν φύγει η κυρία. Αν έχετε κάτι να συζητήσετε έξω παρακαλώ. Thank you. Uh, the first question is to Jean-Paul Σας ευχαριστώ. Jean Paul Gauzès για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάνατε δηλώσεις πολύ γενικές, κύριε Κωνσταντσο. Έχω όμως εγώ πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση. Πώ ε, κρίνεται τι δράσει τη Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τη διάρκεια τη κρίση που δυστυχώ ε, δεν έχει ακόμη τελειώσει. Δεύτερον, η ε, αρχιτεκτονική τη επιτήρηση, και ασφαλώ θα γνωρίζετε ότι υπάρχει απόκληση μεταξύ Συμβουλίου, ΕΚΟΦΗΝ και Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα τη δική σας θέση. Και εν τέλει, μιλήσατε για τους ε, οργανισμούς Πώ πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Ξέρετε ότι αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ε, βλέπω ότι όταν ε, κρίνει ο κόσμος αυτό που κάνουμε, η κρίση που εκφράζεται είναι πάντοτε θετική και μάλιστα από σχολιαστές που συχνά είναι ακόμη και αρνητικοί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακούμε πάντα σχόλια θετικά αυτόν τον καιρό. Αυτό που μπορεί να, πια, να πράξει άλλωστε μέσα σε τέτοιες συνθήκες μια κεντρική τράπεζα είναι ε, είτε να δώσει ρευστότητα στη χρηματοπιστωτική αγορά για να τη βοηθήσει να ε, αντιμετωπίσει την κατάσταση, την κρίση, ιδιαίτερα στην νομισματική αγορά που δεν λειτουργεί πια, όπως ξέρετε, και το... κατά τρόπο μάλιστα πολύ δραστήριο, θα έλεγα επιθετικό σχεδόν. Και το δεύτερο, να αλλάξει η νομισματική πολιτική. Και αυτό επίσης το πράξαμε από τη στιγμή που οι Lehman Brothers κήρυξαν πτώχευση. Εκεί που φάνηκε δηλαδή ότι θα περάσουμε σε ύφεση και ότι κίνδυνος πληθωρισμού δεν υπήρχε. Επομένω δεν υπήρχε κίνδυνος να χάσουμε τον πρώτο στόχο που ορίζει η συνθήκη. Και έτσι με επίσης επιθετικό τρόπο προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίξει στο βαθμό που μπορούσε την οικονομία έναντι του κινδύνου της ύφεσης, των κινδύνων της ύφεσης που εμφανίστηκαν. Το πρέπει να κάνει μια κεντρική τράπεζα, αυτό πράξαμε. Και θεωρώ ότι το πράξαμε με απόλυτα επαρκή τρόπο το πρόβλημα της οργάνωσης των θεσμικών οργάνων, τα θεσμικά ζητήματα. Το κάλυψα στις απαντήσεις μου στο ερωτηματολόγιο, όπως και σήμερα στην παρέμβασή μου. Δηλαδή θεωρώ ότι εν γέννη συμφωνώ με την οργάνωση που έχει οριστεί Έχω πει επίσης ε, στη γραπτή μου απάντηση ότι θα πρέπει μακροπρόθεσμα οι τρεις αρχές να μετατραπούν σε δύο, να εξελιχθούν σε δύο. Ένα σύστημα διπλής εχμής, Twin Peaks όπως το ονομάζουμε, το οποίο γενικώ υποστηρίζω. Και δίνω και τα σχετικά στοιχεία στην απάντησή μου. Και επίσης, σε σχέση και με την έκθεση που ετοιμάσαμε για την Επιτροπή σας, έχω δύο παρατηρήσεις διατυπώσει μέσα σε απαντήσεις μου, όπου επισημαίνω και κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα όσα εσείς. Εν τέλει δε, για τους ε, οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης, τελειώνω πρόεδρε, αυτό που θα πρότεινα ως στοιχείο βελτίωση ήταν να αποκλειστεί ο ρόλος τους από κάθε κανονιστική, ρυθμιστική δηλαδή δραστηριότητα. Γιατί μάλιστα τώρα βλέπουμε ότι έχουν και, ε, τους έχει αποδοθεί αξία και με το παραπάνω. Πράγμα το οποίο μας οδηγεί σε λάθη, σε προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να τους αποκλείσουμε τελείως από την ε, ε, από τις ε, ρυθμιστικές μας επιλογές. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, επαρκή έλεγχο και ρύθμιση τους, πράγμα το οποίο δεν είναι δεδομένο καθόλου στην Ευρώπη και δεν υπάρχει και εποπτεία στην Ευρώπη επαρκής. Ευχαριστώ κύριε Σφέιο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να θε... χαιρετήσω τον κύριο Βίτρο Κωνστάσιο και να του θέσω την εξή ερώτηση. Θα ήθελα να αναπτύξετε λίγο περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αναλύσατε την πρόταση για το ιδέσμη εποπτείας στην αρχική σας ε, εισήγηση και στι γραπτές σας ε, ε, απαντήσεις και δηλαδή πώς θα προβλέπετε εσείς την διαδικασία εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πιο συγκεκριμένους όρους και ήθελα να γνωρίζω δηλαδή ποιον ρόλο θα πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο πλαίσιο των όσων καθορίζουν τα ε, διάφορα ε, καταστατικά σας όσον αφορά την μακροπροληπτική ε, δραστηριότητα και πώς θα μπορέσει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διαρθρώσει τις δράσεις της ε, με τέτοιο τρόπο και να τις συντονίσει με τις νέες αρχές εποπτείας στο ευρωπαϊκό επίπεδο που πολύ πιθανότατα θα έχουν ε, επίσης εξουσίες και αρμοδιότητες σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ κύριε Φέιο, για την ερώτησή σας και αν δεν σας πειράζει θα απαντήσω στα αγγλικά γιατί πιστεύω ότι είναι ευκολότερο για όλους. Φυσικά θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να σας απαντήσω στα πορτογαλικά, όπως θα φαντάζεστε. Answers ε, Όσον αφορά λοιπόν τις απαντήσεις στην ε, εισηγητική μου, στην, στην εισήγησή μου μάλλον, ε, μιλάτε για τη ε, ρύθμιση αυτή και τη νέα αρχή που ορίζεται για την εποπτεία και την ρύθμιση στην Ευρώπη. Είμαι θετικός ως προς αυτό και έχω μελλοντική, μια, μια άποψη όσον αφορά τις δύο αρχές, δηλαδή τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα. Πιστεύω πως από θα πρέπει να εξετάζονται οι δύο αυτοί γιατί ε, τη σήμερα ημέρα υπάρχει διασύνδεση τόσο στενή αυτών των δύο τομέων για τα προϊόντα που πολλούν ε, ε είναι ευρύτατα Και μάλιστα πολλοί από τους ευρωπαϊκούς ομίλους έχουν δραστηριότητες και στους δυο τομείς και για, αυτούς, για πολλούς λοιπόν και διάφορους λόγους πιστεύω πως από κοινού θα πρέπει να εξετάζονται και τα χρεόγραφα να είναι χωριστά οι τίτλοι. Ε, τα μοντέλα που έχουμε μέχρι τώρα δεν λειτουργήσαν καλά κατά τη διάρκεια της κρίσης γιατί υπάρχει διαφορά προσέγγισης ανάμεσα στα δύο πράγματα. Όσον αφορά την εποπτεία δηλαδή του τραπεζικού και του ασφαλιστικού τομέα, το βασικό ενδιαφέρον ε, αφορά ε, στην ανάλυση και προστασία των θεσμών ε, ότι αυτό είναι το βασικό δημόσιο συμφέρον, δηλαδή η προστασία των καταθετών και των, στην περίπτωση των τραπεζών και των πελατών στην περίπτωση των ασφαλιστικών εταιριών. Ενώ στη, ε, τα μία τίτλων είναι εκεί η προστασία των επενδυτών, των ε, μετόχων. Εντάξει, αλλά είναι δύο διαφορετικές ε, προοπτικές και πιστεύω πως η, ο διαχωρισμός των δύο είναι απαραίτητος. Επίσης, η σύνδεση τράπεζας, τραπεζικού τομέα και ασφαλιστικού είναι σημαντική με την, τον αποκλεισμό του, τομέα των τραπεζικών, των, κεντρικών τραπεζών που θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο με τις υποπτικές αρχές της κάθε χώρας. Τώρα, όσον αφορά το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό όπως είπα, μπορεί να λειτουργήσει καλά γιατί στην σύνθεσή του υπάρχει η Κομισιόν αλλά και η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Οργάνου. Όλοι είναι παρόντες δηλαδή, τόσο οι κεντρικοί τραπεζίτες που είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση της κατάστασης και να εκδίδουν προειδοποιήσεις ε, και συστάσεις, αλλά και αυτοί που υποτίθεται πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις είναι παρόντες στο ίδιο Συμβούλιο, άρα μπορεί και να λειτουργήσει. Ωστόσο, ωστόσο, εξακολουθώ να έχω και κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με τα μέσα που δίνονται σε ένα τέτοιο οργανισμό και το ίδιο βέβαια ισχύει και σε άλλες χώρες. Αυτή η λειτουργία επίσης εξετάζεται στη ΣΥΠΑ. Ε, δεν δίνει στον οργανισμό μακροπροληπτικής ε, εποπτείας αρκεπαρκή μέσα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και ίσω λοιπόν σε αυτό το σημείο θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια τελική παρατήρηση. Α, με βάση τη συνθήκη η ΕΚΤ δεν έχει κανένα εποπτικό ρόλο. Και ιδιαίτερα στην προληπτική εποπτεία. Υπάρχει και συγκεκριμένο άρθρο που τα λέει αυτά. Μόνο μια ομόφωνη ψηφοφορία από το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τέτοιο ρόλο στην ε, τράπεζα ή κομμάτι του ρόλου στην ΕΚΤ. Α, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν η ΕΚΤ δεν έχει τέτοιου λειτουργία. Και επιπλέον, μην συγχαίρετε παρακαλώ την λειτουργία του Ταμείου ε, Συστημικού του Συμβουλίου μάλλον Συστημικού Κινδύνου με την ΕΚΤ. Εμείς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία αυτού του νέου οργανισμού, αλλά είναι ένας νέος οργανισμός με δικό του, δική του νομική, νομικό πρόσωπο και δεν ε, εμπίπτει στη λειτουργία και στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ε, γνωμισματική πολιτική, αλλά δεν θα είναι είναι ε, και, το, και το, το Συμβούλιο αυτό δεν θα είναι υπεύθυνο για την οικονομική σταθερότητα ή τίποτα άλλο, μόνο για την εποπτεία. Λοιπόν, παρακαλώ να περιορίσετε τις απαντήσεις σας εντός των 3,5 λεπτών, παρακαλώ. Και γιατί οι υπόλοιποι βουλευτές δεν θα μπορούν να πάρουν το λόγο τότε. Η κυρία Λούλινγκ είναι η επόμενη μιλήτρια από πλευρά του ΕΛΚ. Επειδή ο κύριος Μαργάγιο δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Οδικητά, πρέπει να σας πω ότι από λογισμό σας όσον αφορά την προεδρία σας στην Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας, ε, ομόφωνα λίγο πολύ μας φέρνει εναντίον σας. Αν δει κανεί τα άρθρα τα οποία δημοσιεύτηκαν από τότε που οριστήκατε από το Συμβούλιο Υπουργών, εγώ βέβαια πρέπει εδώ να πω ότι πρόκειται για τον αγγλικό, τον γαλλικό, τον γερμανικό τύπο, ο οποίος εκφράζει μεγάλες επικρίσεις όσον αφορά τη δράση σας. Επικρίσεις που δεν έχει να κάνει με πολιτικούς ε, προσανατολισμούς, είναι επικρίσεις που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες κατέστρεψαν πολλούς αποταμιευτές εξαιτίας ε, της δικιάς σας ε, ελαφρότητας στην κρίση σας. Λοιπόν, κύριε Δικητά, τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τις αποταμιεύσεις τους την περίπτωση της εθνικοποίησης της ΜΠΕΛ. Τι έχετε να πείτε για την BPP, όπου και εκεί η τράπεζα δηλαδή της Πορτογαλίας δεν έκανε τη δουλειά της ό,τι έπρεπε. Και υπάρχει και η Μπέσεπε. Λοιπόν, είναι τρεις περιπτώσεις πολύ σημαντικές. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ για έναν άνθρωπο. Καταλαβαίνω βέβαια το ότι πολλοί δικοί σας χαίρονται να σας βλέπουν εδώ υποψήφιο γιατί νιώθουν ότι σας ξεφορτώνονται κατά κάποιο τρόπο. Αλλά εγώ δεν χαίρομαι, μήπω μπορείτε να μας πείτε πώς κάποιος ο οποίο απέτυχε στη χώρα του μπορεί τώρα να υποστηρίξει ότι μπορεί να αναλάβει την εποπτεία στην Ευρώπη. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την προοπτική. Βλέπετε είναι σαν ε, να δίναμε σε έναν πυρομανή τα μέσα για να βάλει φωτιά. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Εμένα δεν με καθησυχάζει καθόλου όλη αυτή η ιστορία. Oui, euh, madame, euh, je, tout d'abord, euh, je peux vous envoyer des... Μπορώ να σας στείλω και ένα σωρό άρθρα από τον τύπο εκατοντάδες που μιλάνε υπέρ των δικών μου δράσεων από τη θέση του διοικητή της ε, Τράπεζας της Πορτογαλίας. Εσείς αναφέρατε κάποιες περιπτώσεις τις οποίες και θα σχολιάσω. Άκουσα πολλά θετικά για τον ρόλο που έπαιξα προστατεύοντας την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική όπως έπρεπε να είναι στην Πορτογαλία. Εγώ τα έβαλα με πολλές κυβερνήσεις και με αυτήν που με όρισε στην τράπεζα για την δικιά της επεκτατική πολιτική που υιοθετήθηκε στην Πορτογαλία. Και το έκανα αυτό στο όνομα των αρχών που απαιτούνται για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής ε, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτά που είπατε εσείς έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες περιπτώσεις που συνέβησαν στο τραπεζικό σύστημα. Γενικά όμως μιλώντας για το τραπεζικό σύστημα, ευχαρίστως να σας στείλω και την ε, αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα της Πορτογαλίας ανέλαβε την εποπτεία του συστήματος στο σύνολό του και απέφυγε με αυτόν τον τρόπο προβλήματα ρευστότητας ή προβλήματα φερεγγιότητας του δικού μας τραπεζικού συστήματος. Αντισταθήκαμε με πολύ θετικό τρόπο στην κρίση και δεν έχουμε προβλήματα στο τραπεζικό μας σύστημα όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι πολύ θετικό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα της Πορτογαλίας ηγήθηκε της ρύθμισης και της εποπτείας των τραπεζών. Έχουμε τρεις περιπτώσεις απατών στο σύστημα το τραπεζικό της Πορτογαλίας. Πρόκειται για απάτες οι οποίες έγιναν σε πολύ ψηλό επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση των τριών αυτών τραπεζών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι φορείς που έχουν εμπειρία σε τέτοια θέματα εποπτείας ποτέ δεν επέκριναν την Τράπεζα της Πορτογαλίας που δεν μπόρεσε πιο νωρί να εντοπίσει τις απάτες αυτές ε, οι οποίες έγινονται. Όπως ξέρετε, οι απάτες που έγιναν σε πολύ υψηλό επίπεδο των ε, τραπεζών αυτών είναι περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν μέσω της εποπτείας. Προσωπικά μιλώντας, επίσης πρέπει να σας πω ότι ω διοικητή τη Τράπεζα της Πορτογαλίας δεν ήμουν άμεσα υπεύθυνο για την εποπτεία. Δεν παρακολουθούσα σε καθημερινή βάση τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες ε, προέβαιναν στην εποπτεία αυτή. Είπα όμω στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο ότι φυσικά και έχω την ευθύνη για όλα όσα γίνονται από την τράπεζα και δεν μετανιώνω για καμία από τις δράσεις που ανέλαβαν οι υπηρεσίες, διότι ήταν αδύνατον να εντοπιστούν τα προβλήματα αυτά. Αυτό το οποίο συνέβη στην BSP, την Κεντρική Τράπεζα, δεν ε, ήταν ε, διάστασης που έθετε σε κίνδυνο την, ε, ή το ίδιο το σύστημα. Ήταν μια απάτη. Δεν δημιούργησε όμως πρόβλημα σε ένα θεσμό ο οποίος ε, πάντα λειτουργεί καλά και στέρεα. Αυτό που συνέβη στην ε, Μπεμέν είναι μία μαζική απάτη. Και ειλικρινά θλίβομαι που δίνεται την ευθύνη στην εποπτεία και όχι στην ίδια την τράπεζα και τους τραπεζίτες οι οποίοι έκαναν εγκλήματα. Μα η υποπτία δεν είναι αστυνομική αρχή. Δεν έχουμε τα μέσα που έχει αστυνομία για να εντοπίζουμε τις απάτες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Όσον αφορά τώρα την ΜΠΠ, η απάτη έγινε στα προϊόντα των κεφαλαιακών αγορών, πράγμα το οποίο δεν είναι ευθύνη της Τράπεζας της Πορτογαλίας. Εμείς δεν έχουμε την εποπτεία αυτών των προϊόντων. Είναι προϊόντα που δημιούργησαν προβλήματα στην ΠΕΡΕΠΕ προϊόντα τα οποία, οικονομικά βέβαια προϊόντα, που είναι ευθύνη άλλης αρχής εποπτείας. Πράγμα που σημαίνει, εντάξει δεν έχω τώρα το χρόνο να σας εξηγήσω τα πάντα, όμως είναι άλλη εποπτική αρχή υπεύθυνη. Η τράπεζα της Πορτογαλίας δεν ευθύνεται και δεν ούτε και αρχή εξάλλου, η εποπτική γιατί όπως σας είπα ήταν δύσκολος ο τοπισμός των απατών αυτών. Πάντως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα της Πορτογαλίας δεν ευθύνεται και εγώ είμαι περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο ε, έφερα σε πέρα στα καθήκοντά μου σε όλο αυτό το διάστημα. Πρόεδρος. Ναι, δεν σας διακόψα γιατί ήταν σημαντικό να απαντήσετε. Λυπάμαι όμως που πρέπει να σας σταματήσω τώρα. Ούργμαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν διατυπώσω την ερώτησή μου, θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Κωνστανσιο, το εξή. Είναι η δεύτερη φορά που έχω την ευκαιρία να σας ακούσω. Γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι ως συντονιστές έχουμε ήδη την, είχαμε ήδη την ευκαιρία να αναπτύξουμε ενδιαφέροντα διάλογο με όλους τους υποψηφίους πριν λάβουμε την απόφαση. Η παρατήρηση μου λοιπόν είναι ότι μας μιλάτε με τρόπο ε, συγκεκριμένο, μας δίνετε στοιχεία, δεδομένα. Εκτιμώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν προσπαθείτε να καλυφθείτε πίσω από ένα διπλωματικό ύφο το οποίο ε, θα σήμερα δεν θα καταλαβαίνει κανείς τι εννοείται. Μου αρέσει που μιλάτε με συγκεκριμένα πράγματα απτά, μετρημένα, σας καταλαβαίνουμε και μας καταλαβαίνετε. Η ερώτηση λοιπόν είναι η Έχουμε βέβαια μια άνευ προηγουμένου κατάσταση με περιβολικό ε, δημόσιο χρέος σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη και ρωτώ πώς θα αποφύγουμε το φαύλο κύκλο Δηλαδή, προσπαθώντας να ε, ξεφύγουμε από την κρίση, να ε, επιβαρύνουμε σε βαθμό αναπηρία σχεδόν την ανάπτυξή μας, έτσι ώστε να μην μπορεί... Και παρακαλώ, Πρόεδρε, θέλω τον ίδιο χρόνο με την Άστριντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι ώστε λοιπόν... Όχι, θα μου φτάσει, θα μου φτάσει. Προσπαθώ να μπω στην ουσία του πράγματος. Έτσι ώστε να μην παρακολύσουμε την ανάπτυξή μας. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν αυτό το φαύλο κύκλο και πώς θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να βγουν από το δημόσιο χρέος, να ξεφύγουν από το δημόσιο χρέος και σε δύο αναλυτικού χαρακτήρα προβλήματα που έχω υπόψη μου θα ήθελα να απαντήσετε. Έχουμε έναν οικονομικό κύκλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή πολλαπλές δομές, περίπλοκες δομές, με διαφορετικούς οικονομικούς κύκλους, ανάλογα με μια διαφορετική περιοδικότητα ανά κράτος μέλος και πώς ε, τους ε, δημοσιονομικούς κύκλους του δανεισμού ενεργητικού ή παθητικού μπορούμε να το συγκρίνουμε με όλα αυτά. Απάντηση, ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τους κινδύνους που αναφέρεται η δυνατότητα ε, των ε, στρατηγικών κρίση, ε, διαφυγής από την κρίση μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ανάκαμψη, το είπατε κι εσείς. Ναι. Θα ήθελα να επισημάνω ωστόσο ότι οι δέσμες που εφαρμόζονται στην Ευρώπη έχουν να κάνουν με το 1,5% περίπου του ΑΕΠ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι τεράστια τα μέτρα Βέβαια αυτά πάνω από τους αυτόματους σταθεροποιητές που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και που οδήγησαν σε μεγαλύτερο έλλειμμα, όπως άλλωστε αναμενόταν ε, σε σοβαρή, κρίση όπως αυτή που είχαμε τώρα. Όμως η, τα κονδύλια, τα ποσά που διατίθενται πάνω από τους αυτόματους ε, ε, προσαρμοστές, σταθεροποιητές δεν ήταν τεράστια. δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν θα μας ξαναρίξουν σε βαθύτερη κρίση, δηλαδή, όπως την, ε, δεν θα παρεμποδίσουν την ανάπτυξη. Και πιο σημαντικό ακόμη αποδεικνύεται να υποστηριχθεί, τον υποστηριχθεί η νομισματική, για να υποστηριχθεί μάλλον η οικονομική δραστηριότητα, αποδεικνύεται ότι ήταν πιο σημαντική η νομισματική πολιτική, δηλαδή η μείωση των επιτοκίων που για τους χρεωμένους οικονομικούς ε, παράγοντες σήμαιναν σημαντική μείωση του κόστους και για τις οικογένειες, για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις που μπόρεσαν να διατηρήσουν ένα επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας ε, αρκετά ικανοποιητικό χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Όσο έχουμε ύφεση βέβαια δεν υπάρχει κίνδυνος ε, πληθωρισμού στο εγγύς μέλλον και μπορούμε να, να, συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε αυτό το ρόλο, να υποστηρίζουμε δηλαδή την οικονομία περισσότερο. Η στρατηγική εξόδου, διεξόδου που υιοθετούμε για την ε, μείωση των επιπέδων ε, το, της στήριξη ρευστό. Της, το μειώνουμε το ρευστό διότι δεν χρειάζεται περισσότερο. Σταθεροποιείται η αγορά σε επαρκές επίπεδο και έτσι η στήριξη σε ρευστό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι πια τόσο απαραίτητη όσο στο παρελθόν ήταν παγωμένες οι αγορές. Τώρα πια δεν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση ε, της ε, δισκαμψίας μπορούμε να προχωρήσουμε δηλαδή περαιτέρω σε μείωση του, της διάθεσης ρευστού. Για την άλλη ερώτηση, για τις σχέσεις μεταξύ ε, απόψεων, μάλλον κύκλων ε, μέσα, και, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ κρατών μελών. Δεν είναι τόσο διαφορετικά. Αν κοιτάξουμε τα επίδα διάχυσης της ανάπτυξης του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη, με την ε, απόκληση κατά μέσο όρο της ανάπτυξης του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη, μπορούμε να διακρίνουμε μία διάχυση μειούμενη από την αρχή της αγωγής του ευρώ μέχρι και μέχρι τώρα. Δηλαδή υπάρχει καλύτερο συγχρονισμός τώρα από ό,τι στην αρχή της εισαγωγής του ευρώ το 1999. Αντικειμενικό στοιχείο αυτό και πολύ σημαντικό. Δηλαδή δείχνει ότι έχουμε διαφορετικούς βαθμούς αλλά την ίδια λίγο πολύ διακύμανση σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κυρία Φερέιρα. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δικητά, εγώ έχω δύο ερωτήσει. Πρώτη είναι, αν δούμε τι συνέβη τα πρόσφατα έτη, έχουμε πολλά ονόματα. Black Rock, Fannie Mae, Lehman Brothers κλπ. κλπ. Σαφή ε, μηνύματα για τι μεγάλες αναταραχές σε όλες τις αγορές αυτές. Άρα λοιπόν για όλες τις χώρες, και για την Ευρώπη και για τη ΣΥΠΑ, τις βλέπουμε τι ε, αντιπροσώπευε όλα αυτά για τον ε, απλό πολίτη όσον αφορά την συνεισφορά του. Την ερώτηση αυτή έκανε η συνάδελφος από το Λουξεμβούργο, αλλά δεν είχε λάβει υπόψη προηγουμένως τις επιπλοκές οι οποίες έγιναν αισθητές στην αγορά του, ε, του Γιατί ήταν αγορές οι οποίες επηρεάστηκαν ε, και ε, ταράχτηκαν από πολύ σοβαρά τραπεζικά προβλήματα. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες ιδέες λίγο πιο πέρα από αυτά που μας παρουσιάσετε. Δηλαδή, να ξέρουμε, να δούμε πώς μπορεί να παρέμβει η τράπεζα εξάντες, δηλαδή πριν ε, να προκύψουν τα προβλήματα. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που υπάρχουν. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το πώς βλέπετε τις δυνατότητες παρέμβασης, τα triggers σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς μπορούμε εμείς να εγγυηθούμε ότι όταν εκ των προτέρων δεν θα, παρέμβει η Κεντρική Τράπεζα δεν θα υπάρχει ε, σύγκρουση με τις ε, εθνικές ε, κεντρικές τράπεζες που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μετόχων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Όπως ξέρετε ότι είναι γνωστό ότι η δημόσια παρέμβαση ήταν ε, πολύ μεγάλη και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και είναι επίσης γνωστό ότι αν εξετάσουμε όλα τα προγράμματα που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή η παροχή κεφαλαίων, ε, η αγορά των ε, τοξικών προϊόντων και τα λοιπά, τα δάνεια είναι τεράστια ποσά. Και στις δύο περιπτώσεις ανήλθαν στο, σε πάνω από 30% του ΑΕΠ. Δεν δαπανήθηκαν όλα αυτά τα χρήματα και δεν θα χαθούν όλα αυτά τα χρήματα, όχι. Αλλά δεσμεύτηκαν ως ένα δίχτυ ασφαλείας και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πολλά χρήματα. Κάποιος υπολόγισε ότι στην περίπτωση των ΙΠΑ όλα αυτά τα χρήματα είναι περισσότερα από τα όσα δαπάνεσαν οι ΙΠΑ σε όλους τους πολέμους στους οποίους συμμετείχαν. Και όπως σας είπα, δεν θα δαπανηθούν, ούτε θα χαθούν όλα αυτά τα χρήματα. Αλλά δεσμεύτηκαν... Αυτό δείχνει, βέβαια, το μέγεθος των τιμών που φτιάχτηκαν ε, στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα, ξεκινώντας βέβαια από τη ΣΥΠΑ. Να σας πω ότι στην περίπτωση της Πορτογαλίας τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί ήταν το 14% του ΑΕΠ. Αλλά το κράτος δεν θα χάσει ούτε λεπτό γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν ε, οι ενέσεις κεφαλαίου, ούτε η αγορά τοξικών κεφαλαίων έγινε, Ορισμένες ε, τράπεζες ε, θα πληρώσουν τα που ήταν αφαιρέγγες, ε, θα πρέπει να πληρώσουν, να πληρώσει το κράτος, αλλά θα αναλάβει απλώς τα δάνεια. Τα δάνεια θα πληρωθούν από τους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν το κράτος δεν θα χρεωθεί ούτε ε, δεκάρα. Πράγμα το οποίο είναι υπέρ της δικής μας εποπτείας. Εσείς τώρα ρωτήσατε τι μπορεί να γίνει εκ των προτέρων. Και αυτό μπορεί να γίνει είναι αυτό που προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Τα δύο κεντρικότερα θέματα είναι τα εξής κατά την απόψή μου. Πρώτον, ρύθμιση και εποπτεία τη συνολική μόχλευση του, δημοσιο... του χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν υπήρχε πριν. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα ποσοστό βάση για τη μόχλευση. Πράγμα από το οποίο σημαίνει πω ε, μεγάλοι κολοσσοί δεν μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα μόχλευση 40%, 40 φορέ μάλλον το κεφάλαιό του και ούτω καθεξής. Πράγμα το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον ε, πολλαπλασιασμό της κρίσης με αρχή τα ενυπόθηκα δάνεια. Έπειτα, δεν υπήρχαν διεθνείς κανονισμοί όσον αφορά τα, τα, τη ρευστότητα ή την ε, αναντιστοιχεία ρευστότητας ε, για τα κράτη. Σε ορισμένε χώρε υπήρχαν κάποιες προβλέψει, αλλά διεθνώ όχι. Στην περίπτωση τη Northern Rock που αναφέρατε προηγουμένω, για παράδειγμα, ένα, είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα αναντιστοιχία μεταξύ των ληξιπρόθεσμων. Ε, ε, δανείων και ασφαλίσεων. Ε, δηλαδή εμείς ε, με αυτόν τον τρόπο τώρα θα είμαστε σίγουροι πως δεν θα υπάρξει υπερβολική χρηματοδότηση όπως όταν μέχρι τώρα και ήταν η βάση για τη σημερινή κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Μπουζή. Κύριε Μας είπε ο κύριος Ζων Κλωτ Κισκλισέ ότι μπορεί να επανεμφανιστούν ε, σημαντικά προβλήματα αν δεν υπάρχουν σημαντικές προσαρμογές ως προς τις ε, κύριες ε, οικονομίες και τα αιτήματά τους. Το G20 αποφάσισαν ε, υπόσχονται μάλλον να κάνουν ακριβώ το ίδιο, αλλά δεν ξέρω αν θα το επιτύχουν με του όρου που το εννοούμε. Και δεύτερον, η Ευρωζώνη στο τωρινή τη μορφή έχει πιθανότητε επιβίωση, πιστεύετε, αν δεν έχουμε μια πιο αυστηρή οικονομική νομισματική αλλά και φορολογική ε, πολιτική και μια κοινή αγορά εργασίας. Λιγότερο από ένα λεπτό, Πρόεδρε. Sorry. Um, global... Ναι, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Δεν μπόρεσε μέχρι τώρα η G20, να το λύσει. Το επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας που απαιτείται για να επιληθεί το πρόβλημα είναι άνευ προηγουμένου. Δεν έχει όμοιό του στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν. Όντω. όμως θα πρέπει όλοι οι κύριοι φορείς, οι κύριοι παράγοντε να αντιληφθούν τι διακυβεύεται εδώ. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξηγούμε διαρκώ ότι μεγαλύτερε χώρε με μεγαλύτερα μεγαλύτερε ανισορροπίε προ τι δύο κατευθύνσει, πρέπει να επιτελέσουν το καθήκον του. Ιδάλω, όπω είπατε και εσεί, από τα λόγια του Πρόεδρου Τρισέ, ναι, κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε του διοικητού Τρισέ, μάλλον κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε νέε κρίσει και στο μέλλον. Αυτό πια είναι στα χέρια των μεγάλων κρατών. Πρέπει να αντιληφθούν τα ίδια το συμφέρον τους το δικό του συμφέρον είναι να συνεργαστούν μακροπρόθεσμα. Διαφορετικά θα έχουμε όλοι προβλήματα και τα ίδια τα κράτη αυτά, αλλά όλοι μαζί, μεγαλύτερα ακόμα προβλήματα από τώρα. Ευρωζώνη και περισσότερο συντονισμό των πολιτικών, οικονομική, φορολογική πολιτική, ναι, ασφαλώς, υπό τι τρέχουσε συνθήκε, είναι απολύτω απαραίτητο ω προ την λειτουργία του συντονισμού της ε, φορολογικής πολιτικής και της ε, χρηστής λειτουργίας της φορολογικής πολιτικής που δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί σε όλα τα κράτη-μέλη όπως πρέπει. Οι μηχανισμοί δηλαδή του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη θα πρέπει να ενισχυθούν. Χρειάζονται ως εκ τούτου κάποιες αλλαγές στον τομέα αυτών καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης και κυρίως από την ε, πτυχή των δεδομένων είναι απαραίτητη. Είναι λυπηρό ότι μόνο εκ των υστέρων σε πολλές περιπτώσεις είναι ε, σαφές το μέγεθος των προβλημάτων ή είναι ορατή η κατάσταση. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Και την άλλη φορά που ήμουν εδώ πάλι, ανέφερα ότι είχαμε και στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια, το ίδιο πρόβλημα και ήμουν επικεφαλής της Επιτροπής που είχε εκπονήσει μία έκθεση την εποχή εκείνη που έδειξε το πρόβλημα με βάση τα δεδομένα που είχαμε. Πράγμα το οποίο δεν χάιδεψε τα αυτιά της τότε κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει όμως Πανεπιστήμιο Διοίκησης. Ε, ε, μετά όμως θεσπίστηκε ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Στατιστικών, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Κεντρικής Τράπεζας, της ε, κυβέρνησης, έτσι ώστε να ε, γίνεται η μελέτη αυτής, ε, αυτών των συνθήκων με τα σωστά στοιχεία και από τη στιγμή που θεσπίστηκε αυτό το όργανο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ω προ τα στοιχεία μα και την αξιολόγησή του. Είναι σημαντικό να υπάρχει τέτοιο όργανο, κατά την άποψή μου. Και είναι σημαντικό, πιστεύω, οι κεντρικέ τράπεζε να συμμετέχουν. Γιατί έχουν καλέ γνώσει των, των συνθήκων και μπορούν να βοηθήσουν. Το Ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Θα χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο και ελπίζω να μου δώσει την ευκαιρία κάποιο άλλο ομιλητή με ερώτηση αντίστοιχη. Εν συντομία όμω πιστεύω ότι είναι δυνατόν δεν είναι απαραίτητο κατά την απόψή μου για να συσταθεί ένα τέτοιο μέσο να αναθεωρηθεί η συνθήκη. Έχω κάποια επιχειρήματα εν προκειμένου στα οποία δεν μπορώ να επεκταθώ. Απλώς δεν βλέπω τι ρόλο επιπλέον, τι επιπλέον έχει να προσφέρει ένα τέτοιο όργανο, δηλαδή τι σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο θα είχε να προσφέρει. Εάν όμως θεωρούμε ότι μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω, ναι δεν έχω αντίρρηση. Ευχαριστούμε. Θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα σίγουρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρου του συναδέρφου Στρέτσεκ, που έπρεπε να φύγει σήμερα το πρωί, δυστυχώ θέτω την ερώτηση αυτή. Και το λέω γιατί η ερώτηση που ακούγεται από το Ενωμένο Βασίλειο μπορεί να ακουστεί διαφορετικά. Θέλω να μου πείτε για την αύξηση της ασφάλισης όσον αφορά το χρέος από τα κράτη-μέλη, γιατί η παρούσα κρίση έδειξε ότι όταν μιλάμε για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να ξέρουμε ότι μιλάμε και για κυβερνήσει και για κράτη ολόκληρα. Πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για ολόκληρο το συστημικό κίνδυνο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συστημικού Κινδύνου φτιάχνεται αυτή την εποχή και θα έπρεπε να αποφεύγει τέτοιου συστημικού κινδύνου στο μέλλον. Οπότε οι ερωτήσει είναι θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όχι μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και άλλους συστημικούς κινδύνους από ανεύθυνες μακροοικονομικές πολιτικές ή φορολογικές πολιτικές ε, κρατών μελών. Και δεύτερον, τι μηχανισμούς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ελέγξει τέτοιους κινδύνους σε κυβερνητικό επίπεδο, σε επίπεδο χωρών και κυβερνήσεων δηλαδή. Ο υποψήφιος. Ναι, Πρώτα μια γενική παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κάτι διαφορετικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων και δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων. Η δουλειά είναι πολύ τεχνική φυσικά και θα ετοιμάζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να πάρει αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Οπότε έχει νόημα η ερώτηση που βάζετε, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η απάντηση λοιπόν στην πρώτη σας ερώτηση είναι ναι. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Και όσον αφορά την φορολογική πολιτική των χωρών, αλλά και όχι μόνο. Θα, κοιτάμε, θα κοιτάει και την γενική κατάσταση της οικονομίας τους και την δημοσιονομική ισορροπία που υπάρχει στην οικονομία της χώρας σε μερικές περιπτώσεις όταν το χρέος είναι υπερβολικό και το έλλειμμα είναι υπερβολικό, αυτό οφείλεται στη συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα μερικές φορές και όχι μόνο του δημόσιου. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να αναλύουμε ολόκληρη την κατάσταση και οι προειδοποίησεις, οι συστάσεις εφόσον πρέπει να γίνονται, θα γίνονται με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Αυτός είναι ο ρόλος του. Όσον αφορά όμως την προετοιμασία, εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει το προσωπικό της προκειμένου να έχει γραμματεία που θα διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις να προετοιμάζει το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Αυτό θα το κάνουμε. Και όταν έρθει η ώρα, όταν έχουν όλα εγκριθεί, θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Φιλιπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Μ' άρεσε πολύ παράγραφος που είχατε βάλει για τα παράγωγα, για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, όπως επίσης και η τελευταία παράγραφος που δείχνει φιλοδοξία. Ωραία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά αυτό είναι αμφίδρομο, γιατί ο μελλοντικό ε, το μελλοντικό αφεντικό σας, αναφέρθηκε στη σύνθεση των προσαρμογών των φορολογικών, αναφέρθηκε στις δαπάνες επειδή λέει ότι έχει αυξηθεί το μέγεθος του δημόσιου τομέα. Οι πολιτικοί καθορίζουν τελικά την πολιτική δράση. Οπότε θέλω να ξέρω, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώς θα το βλέπει αυτό, πώς θα το ερμηνεύσει αυτό. Γιατί το μέγεθος του δημόσιου τομέα είναι πολιτική απόφαση. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο ιδιωτικό τομέα όπω το Ηνωμένο Βασίλειο ή ο δημόσιο αλλού, αλλά είναι θέμα πολιτική επιλογή. Οπότε το μέγεθο του δημόσιου τομέα για μένα δεν είναι επιχείρημα. Και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ακολουθεί τις, ε, τα καθήκοντά τη, ε, τον ρόλο τη και τίποτα παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ποια είναι η πολιτική σκέψη και αυτό θέλω να ξέρω για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει μία σχολή σκέψης για την ανάπτυξη για παράδειγμα που το χρησιμοποιεί συνέχεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποιοι είναι οι δείκτες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και πιο συγκεκριμένα εσείς τι θα κάνετε μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ε, δώσετε όθηση σε περισσότερες σχολές σκέψης. Τι εννοώ με αυτό. Αν εξαρτάστε από ένα ρεύμα μόνο και υπάρξει εκεί κάποιο πρόβλημα, πεθαίνετε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες. Δεν κατάλαβα. Ρωτώ υποψήφιο. Μιλήσατε για εναλλακτικού δείκτε, εναλλακτικού σε τι. Μα στο ΕΠ, απαντάει ο κύριος Λάμπερτ απάντηση από τον υποψήφιο. Αυτό είναι δύσκολο. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δεν θα ερμηνεύσω εγώ αυτά που είπε ο πρόεδρος Τρισέ, ούτε θα σας πω εγώ τι εννοούσε, γιατί δεν ξέρω τι είπε, οπότε δεν θα σχολιάσω τα όσα σας είπε. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι ποτέ δεν θα με δείτε να κάνω δήλωση όπου να συζητάω το επίπεδο δαπανών στη μία την άλλη χώρα. Και αυτό γιατί αν δείτε την ευρωπαϊκή σκηνή θα διαπιστώσετε ότι εδώ και πολλά χρόνια η Ιρλανδία ήταν μια πολύ ανταγωνιστική οικονομία, ιδιαίτερα επιτυχής και ανταγωνιστική, με πολύ χαμηλό επίπεδο ε, δαπανών. Από την άλλη μεριά έχετε τη Δανία, επίσης πολύ ανταγωνιστική, βάσει των δικτών ανταγωνιστικότητα. ιδιαίτερα επιτυχή λοιπόν, αλλά με εντελώ διαφορετικό επίπεδο δαπανών. Οπότε και οι δύο πέτυχαν και οι δύο ήταν ανταγωνιστικές, οπότε δεν θα με ακούσετε ποτέ να κάνω τέτοιου είδου σχόλια. Εναλλακτικοί δείκτες τώρα. Άλλοι, άλλες σχολές σκέψης. Εγώ είμαι υπέρ του να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε εναλλακτικού δείκτε. Το, έχει κάνει, το έχουν κάνει τα ΗΕ, υπάρχει και εκεί. Είναι κάτι πολύ καλό σαν προσπάθεια. Στη Γαλλία υπήρξε πρωτοβουλία από τον πρόεδρο Σαρκοζή να δημιουργήσει μια επιτροπή που να το εξετάσει. Και εγώ, ναι, ευχαρίστως. Αν υπάρχουν νέοι δείκτες αποδεκτοί, σε διεθνέ επίπεδο αν υπάρξει μια τέτοια αλλαγή, τότε ναι, βεβαίω θα μπορούσαμε και εμεί να χρησιμοποιήσουμε τέτοιους εναλλακτικού δείκτε. Αλλιώ δεν είναι ο δικός μας ρόλος να αποκλίνουμε από τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας και που είναι σημαντικά προκειμένου να αξιολογήσουμε τους κινδύνους πληθωρισμού. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε τώρα. Ευχαριστώ, λέει πορτοκαλικά ο Ο κύριος Πόσταρ τώρα. Πόρτας. Πόρτας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βίκτορ Κωνστάσιο, θέλω να σας υποβάλω ερωτήσεις όσο γίνεται πιο ξεκάθαρες, ώστε αυτές να εξαρτηθεί και η ψήφος μου. Καταρχήν, ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση των ε, οργανισμών βαθμολόγησης ή επιστολεπτικής αξιολόγησης, είτε να, να ανεξαρτοποιηθούν αυτές οι τέσσερις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε να δημιουργηθεί μια νέα ευρωπαϊκή, ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης. Θέλω να έχω την άποψή σας. Και η άλλη άποψη που θα ήθελα να ακούσω είναι κάτι που για μένα είναι προφανές. Η άνηση κατανομή των θυσιών με βάση τα διάφορα σύμφωνα σταθερότητα και ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό και σας ερωτώ, σε θέματα offshore, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με παγκόσμια ρύθμιση, είτε και με το τέλος αυτών των παραδείσων ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά για το τι θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη όσον αφορά μάλλον τι θα γίνει στην Ευρώπη, όσο αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν. Ε, αν είστε δηλαδή όχι στην εφαρμογή πολύ αυστηρών ε, κανόνων και φόρων για με, τα εμβάσματα που γίνονται προς τους φορολογικούς παραδείσους από την Ευρώπη. Και έπειτα τα ευρωομόλογα να σας ρωτήσω για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ή τα ευρωομόλογα, γιατί στη θεωρία αυτά μπορούν να απορροφήσουν κομμάτι των, ε, κρατών, των χρεών των κρατών και μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τα έσοδα τα αντίστοιχα. Γιατί λοιπόν να μην το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σοβαρά την περίπτωση έκδοση ευρωομολόγων. Και ένα σύντομο σχόλιο και μια παρατήρηση για τον ε, κύριο Βίτορ Κωνστάνσιο για το ότι, έκαν, για το ότι το πορτογαλικό κράτος να χάσει ούτε ένα ευρώ με το τραπεζικό πρόβλημα. Ναι, δεν έχασε αλλά η, το, από τα, το της Πορτογαλίας έχασε αρκετά. Ο υποψήφιο αυτό δεν έχει να κάνει με την κρίση, με τα προγράμματα που φτιάξαμε για να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα και η Κάισα Ζεράλ ε, δεν θα χάσει ούτε λεπτό είπαμε γιατί το κράτος το στηρίζει και θα <coughs> κεφαλαιοποιήσει αν αυτό χρειαστεί. Δεν έχει αυτό να κάνει λοιπόν με το κρίση και το τραπεζικό τομέα γενικότερα. Τώρα σε σχέση με τους οργανισμούς αξιολόγησης ε, φυσικά αυτό που είπα είναι ότι είναι πιστεύω σημαντικό οι βαθμολογήσεις από τους οργανισμούς αυτούς να μην παίξουν ρόλο στο επίσημο ρυθμιστικό σύστημα και είναι δυνατόν να απευθυνθεί κάτι τέτοιο χωρίς να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε νέο οργανισμό. Οι οργανισμοί που υπάρχουν θα συνεχίσουν να λειτουργούν, η αγορά θα τις λαμβάνει υπόψη ή όχι, όπως ε, θεωρεί σωστό, αλλά μπορεί να αποφύγουμε την χρήση των αξιολογήσεων για επίσημους ρυθμιστικούς σκοπούς. Και αυτό είπα, πέρα από την υπόθεση της καταγράφησης, της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του ΣΥΝ, πράγμα το οποίο δεν γίνεται ακόμα, να λυθούν πραγματικά πιθανέ συγκρούσει συμφερόντων ανάμεσα στο ρόλο του ω οργανισμού αξιολόγηση και το ρόλο του ως συμβουλευτικών σωμάτων ή οργανισμών. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν λοιπόν, αλλά η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού η δημιουργια ενο αυτή καθ' αυτή δεν θα άλλαζε το κατάσταση, το τοπίο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το ρυθμιστικό σύστημα να έχει τις δικές του μεθόδους και τα δικά του ε, μέσα και δείκτες. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, που βασικά αφορούσε τους ε, φορολογικούς παραδείσους, να σας ε, παραπέμψω σε μια από τις απαντήσεις που έδωσα στο ερωτηματολόγιο, όπου Μία σελίδα έγραψα αντιμετωπίζοντα και μάλλον αναλύοντα το θέμα των παραδείσων. Δεν είναι αλήθεια πω δεν έχει γίνει τίποτα διεθνώ. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των ταμείων, των φόρων δηλαδή και των εσόδων ε, πολλών χωρών. Τώρα δηλαδή οι παράδεισοι πρέπει να συμμορφούνται προ κανόνε που παλιότερα δεν υπήρχαν καν. Τώρα, Όσον αφορά τις ε, εποπτικές λειτουργίες πρέπει να γίνουν περισσότερα, διότι σε ορισμένους παραδείσους, ας πούμε, δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόσβαση στον τελικό δικαιούχο για το οποίο θέμα πολλές φορές ε, δεν μπορεί να υπάρξει και υποπτία μάλλον λόγω αυτού δεν μπορεί να υπάρξει και υποπτία. Αυτό χρειάζεται να γίνει μετά την κρίση. Τώρα για τα ευρωομόλογα, η ΕΚΤ δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα. Στην, ε, δεν συμμετέχει η ΕΚΤ στην έκδοση ευρωομολόγων. Το να συμμετέχει στην έκδοση ομολόγων κάποιου κυρίαρχου κράτου θα ήταν κατά τι συνθήκε, γιατί το άρθρο 3 νομίζω λέει σαφώ πω η Ένωση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν μπορεί να αναλάβει χρέο από άλλε χώρε ή από κάποιο δημόσιο ε, οργανισμό. Αν υπήρχε τέτοιο ρόλο λοιπόν για τα ευρωομόλογα θα ήταν με διαφορετικό τρόπο και όχι να απορροφήσουν το χρέο των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Godfrey Bloom. συγγνώμη, όλο κάνω λάθος, λέω Jeffrey αντί για Godfrey. Μην ανησυχείς και όλοι μου συγγενείς το ίδιο κάνουν. Θα ήθελα να πω ε, ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Από οικονομική πτυχή, και το λέω αυτός οικονομολόγος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κατασκευασμένη ως μια νομισματική ζώνη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, να επιβιώσει μακροπρόθεσμα εάν δεν έχει δημοσιονομική πειθαρχία ή κάποια πολιτική, εν περιπτώσει, με βάση την οποία ένα είναι αυτό που θα έχει την ευθύνη τη χάραξη φορολογική πολιτική για τα κράτη-μέλη. Όταν υπάρχει δυνατότητα μεταφορά κεφαλαίων, τη στιγμή που έχουμε χώρε όπω η Ελλάδα που εκδίδουν τα δικά του ομόλογα, έχουν μειωθεί τα spread και αυτό σημαίνει μόνο ότι παρατείνεται η διάρκεια του χρέους και εξάγεται το πρόβλημα. Ποια είναι η άποψη σας προκειμένου. Απάντηση. Ευχαρίστως να απαντήσω. Θα χρειαστώ όμως περισσότερο χρόνο για να, ικανοποιήσω, για να απαντήσω πλήρως στα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θέτεται. Εν πάση περιπτώσει όμως να κάνω ένα σχόλιο για τους νομισματικούς χώρους. Ίσως υπάρχει μια σύγχυση, ίσως επικρατεί σύγχυση προς το τι εννοεί ως ultimate currency areas η οικονομική θεωρία. η θεωρία αυτή δεν θεωρεί ότι για να έχουν οικονομική ενό... ένωση χρειάζεται να έχουν το ίδιο επίπεδο δραστηριότητα ή ανάπτυξη. Η οικονομική θεωρία ερευνά μόνο και προσδιορίζει κριτήρια. για τα εναλλακτικά ως προς, το, ε, ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μέτρα Τα μέτρα δηλαδή αυτά που θα εξασφαλίσουν την προσαρμογή της ε, οικονομίας τους κλειδονισμούς και τις ανισορροπίες. Και αν δείτε τον Ρόμπερτ Μαντέρ που ήταν ο πρώτος ο οποίος μελέτησε τις τιμές και, τους, και τις αμοιβέ, αφενός και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαντήσεις με τον Πίτερ Κάνον ο οποίος λέει εναλλακτικέ στους ασυμμετρικούς κλειδονισμούς είναι η διαφοροποίηση μιας χώρας, μια παραγωγική δομή δηλαδή διαφοροποιημένη και όχι επικεντρωμένη σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Και ο μακίναν λέει, σημαντικό είναι αν η χώρα μικρή και πολύ ολοκληρωμένη, πολύ ενοποιημένη δηλαδή, ε, νομισματικά, μέσα στην ονομασματική ένωση δούμε πως η ε, οικονομική ολοκλήρωση μέσα στην Ένωση θα στηρίξει αυτήν ε, την θεωρία. Αυτά είναι, ε, αυτές είναι οι θεωρίες στο τομέα της νομισματικής, στο νομισματικό μάλλον τομέα. Αυτό που γίνεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρωζώνη, είναι ότι υπάρχει μεγάλη ολοκλήρωση έπειτα. είμαστε δεσμευμένοι σε ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και μέσα σε αυτές τις συγκεκριμένες περιστάσεις για μια μικρή οικονομία να μπει στο ευρώ είναι πολύ πολύ πλεονεκτικό. Πολύ, για μια μικρή οικονομία με ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και με πολύ ολοκληρωμένη οικονομία η συναγχρηματική ισονοτιμία δεν παίζει ρόλο γιατί αν η αλλαγή χρησιμοποιείται, μάλλον αν η ισοτιμία είναι στην αξία τότε το πραγματικό, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δεν μπορεί να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Μια τέτοια χώρα να αποκομίσει τα ωφέλη τη, τη, του κόστους ε, των ε, συναλλαγών για να χάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία δεν είναι και τόσο μεγάλο κόστος. Υπάρχει δηλαδή μια λανθασμένη αντίληψη ότι δηλαδή μια περιοχή βέλτιστου νομίσματος θα πρέπει να αποτελείται από μια περιοχή με ισότιμες ε, χώρες όσον αφορά την ανάπτυξή τους. Όχι το επίπεδο ε, εισοδημάτων ε, αλλά και ημερομισθείων ε, θα πρέπει να συνδέεται με το επίπεδο παραγωγικότητας της συγκεκριμένης οικονομίας και γι' αυτό και η επιτυχή στη συμμετοχή στην Νομισματική Ένωση βασίζεται σε δύο, τομείς, σε δύο σημεία από μακροοικονομικής άποψης. Πρώτον, τον λαμβάνονται υπόψη οι ανεξελίξεις στο κόστος της μονάδας αλλά και να υπάρχει η παρακολούθηση των αντικυκλικών ε, ε, σημάτων, γιατί αυτό είναι μόνος, η μόνη λύση που έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα έναν ε, γύρο με μια πολιτική ομάδα που έχει το δικαίωμα να φέρει έσταση, αλλά θα πρέπει όλοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, οπότε τώρα οι πράσινες και οι κίτρινες κάρτες θα χρησιμοποιηθούν. Επόμενος ομιλητή είναι ο Ότμαρ Κάρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρωί. Πρώτη παρατήρηση. Χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε την ευκαιρία να σα δούμε για δεύτερη φορά και να συζητήσουμε μαζί σα. Και αυτό όχι μόνο γιατί έχουμε να σας κρίνουμε, αλλά και να μπορούμε και να συγκρίνουμε. Ήταν καλό το ότι δεν είχαμε την υποχρέωση να δώσουμε τον ορισμό αμέσως μετά την πρώτη ακρόαση και ότι έχουμε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στο εξή. Είπατε μόλις τώρα ότι δεν θα σχολιάζατε ποτέ το ύψος των εσόδων ενός κράτους μέλους. Ελπίζω να σας κατάλαβα λάθος, γιατί αν κάποιο κράτος μέλος ε, παραβιάζει του όρου του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, θα πρέπει να τοποθετήσετε. Δεύτερον, μίλησατε για το νομισματικό ταμείο λέγοντας ότι δεν γνωρίζετε τι χρειάζεται κάποιος όταν ακόμη δεν είναι, γνωστά, όταν δεν είναι γνωστό τι μπορεί να κάνει. Ερωτώ λοιπόν, γιατί έχει η Ελλάδα πρόβλημα εάν το ζήτημα είναι τα λεφτά, τα χρήματα, γιατί δεν πάει στο νομισματικό ταμείο να τα ζητήσει. Επίσης, είπατε ότι δεν έχει καθήκον επιτήρηση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ερωτώ, είστε υπέρ μιας ευρωπαϊκής επιτήρησης. Επιτήρηση που θα σημαίνει ότι αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός θα έχει και τον τελευταίο λόγο εάν δεν συμφωνεί μαζί του η Εθνική Αρχή Επιτήρησης απάντηση. Για την πρώτη σας ερώτηση, ίσως δεν με καταλάβατε καλά, διότι αυτό που είπα είναι δεν σχολιάζω το επίπεδο αυτό αυτό. Άλλο είναι να πω εκτιμώ την κατάσταση των δημοσιονομικών μιας χώρας, ιδιαίτερα το έλλειμμα, το επίπεδο του χρέους. Εάν μια χώρα έχει υπερβολικό έλλειμμα, και υπερβολικό επίπεδο χρέου, ασφαλώ και είμαι υποχρεωμένο να τοποθετηθώ, όπω άλλωστε έχω πράξει και για τη δική μου την πατρίδα ω διοικητή τη Κεντρική μου Τράπεζα. Αλλά δεν θα σχολιάσω τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν να κάνουν με αυτή την πολιτική. Αυτό είναι το ε, καθήκον της Επιτροπής, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Αυτό πάντοτε το, το προσέχω με ιδιαίτερη ευαισθησία. προς τα υπόλοιπο όμως και το υπερβολικό έλλειμμα έχω επικρίνει και για τη δική μου την πατρίδα και θα συνεχίσω να το πράττω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Απλώς το επίπεδο αυτό καθεαυτό των δαπανών δεν σχολιάζω. Αυτό εννοούσα. Για το, για το νομισματικό ταμείο. Δεν είναι σαφές για μένα τι θα μπορούσε να προσφέρει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Τι επιπλέον δηλαδή Κάτι που δεν θα μπορούσε να έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ε, θεματοφύλακας της σταθερότητας ή η επιτήρηση και ο έλεγχος, η πιέση αν θέλετε από τους ομολόγους, τα, τα, τα κράτη-μέλη δηλαδή προς το κράτος το οποίο έχει τα προβλήματα προκειμένου την Ελλάδα. Αλλά θεωρώ ότι νομικά δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί η συνθήκη για να, για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο όργανο. Μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό μέσω τη ενισχυμένη συνεργασία ω μεθόδου, βέβαια με απόλυτο σεβασμό κάθε άρθρου τη συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου και του υπαριθμών 123 του άρθρου για το λεγόμενο low bailout, δηλαδή την την διέξοδο από την κρίση. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη τι σημαίνει αυτό το bailout. Α, σημαίνει, πάνω απ' όλα πρέπει να επισημάνω ότι απαγορεύεται να λάβει κράτος μέλος, ε, να αναλάβει μάλλον κράτος μέλος ε, χρέος κάποιου άλλου κράτους μέλους μπορεί να μειώσει, μπορεί να δώσει επιδότηση, μπορεί να αναλάβει την... δεν μπορεί να μειώσει, να επιδοτήσει, να αναλάβει μέρος ή ολόκληρο το χρέος κάποιου άλλου κράτους μέλους. ωστόσο η πίστοση δεν είναι bailout, δεν είναι ανάληψη χρέους, είναι κάτι διαφορετικό και εφόσον δεν επιδοτείται, εφόσον έχει φυσιολογικές συνθήκες, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τη λύση του bailout, της σανίδας σωτηρίας γιατί θα πρέπει να καταβάλουν το επιτόκιο οι Έλληνες, όπως κάθε άλλος. Δεν θα έχει δηλαδή ευνοϊκότερες συνθήκες. Θα έχει απλώς μια διευκόλυνση ως προς την βραχυπρόθεσμη ρευστότητα που χρειάζεται. Αυτό θα της προσφέρουμε, τίποτε άλλο. Εάν θεωρηθεί δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα, στα κατάλληλα επίπεδα, στις αρχές δηλαδή του Συμβουλίου που θα λάβουν την απόφαση, ότι χρειάζεται ένας νέος μηχανισμό, ένα μηχανισμό ο οποίος θα μπορέσει, θα προσφέρει ενδεχομένω τέτοιου είδου ε, στήριξη, εγώ δεν θα είχα καμιά αντίρρηση, διότι πιστεύω πιστεύω ότι θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο να επιτευχθεί υπό το ισχύον πλαίσιο. Εφόσον όμως αναγνωρίζετε όπως σας είπα, από τις αρμόδιες αρχές ότι είναι δυνατό αυτό. Γιατί αν δεν το θεωρούν απαραίτητο, δεν ε, θεωρώ ότι υπάρχει άλλο πρόβλημα. Αν χρειαστεί όμω ένα Ευρωπαϊκό Σωματικό Ταμείο, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση τη συνθήκη. Η πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Ε, Υπήρχαν ακόμη δύο ερωτήσεις. Ε, μία αφορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τελευταία λέξη και η άλλη γιατί δεν πάμε στο Διεθνές Νοσηματικό Ταμείο ή το Ευρωπαϊκό Νοσηματικό Ταμείο. Εάν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε όταν ε, ξαναδοθεί ευκαιρία με, τους, με κάποιον άλλο μιλητή. Κυρία Ντατσί εντωμεταξύ. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο παρατηρήσεις μόνο. Εχθές ακόμη εδώ ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έλεγε ότι από κοινού οικοδομούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νομισματική Ένωση και έχουμε να κάνουμε μια κοινότητα πεπρωμένου. Για την κρίση της Ελλάδας, λοιπόν, ερωτώ, πιστεύετε ότι θα πρέπει να δεσμευθεί κάθε, κάποιο κράτος για την ε, υποστήριξη της Ελλάδας. Πέραν ε, των διμερών συμφωνιών υπάρχει ανάγκη για προσφυγή στο Διεθνές Σωματικό Ταμείο, όπως φαίνεται ότι πιστεύει ο κ. Ζων και επιπλέον για το μέλλον της ζώνης του ευρώ και τον τρόπο λειτουργίας της και μάλιστα πάνω απ' όλα την έλλειψη συντονισμού της οικονομικής Πολιτική Ελλάδα δεν ήθελα τι θέσει αυτές για να καταλάβω τι άποψη έχετε και εσεί. και θα ήθελα να ρωτήσω τι ορισμού και τι αντιλήψη έχετε για αυτήν την υπόθεση. τα κατά άλλα Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι... Ε, δεν είναι η κάστα ειδική. Οι βουλευτέ κάνουν σοβαρή δουλειά, αλλά κάνουν και οι βοηθοί του αρκετά σοβαρή δουλειά και πρέπει και αυτού να του σεβόμαστε, όπω και του βουλευτέ κύριος Κωνστάνσιο. Ευχαριστώ πολύ αν μου επιτρέπετε να απαντήσω στα αγγλικά για να είμαι πιο ακριβής και πιο ταχής για το Διεθνές Νοσηματικό Ταμείο. Και εγώ, όπως πιστεύω και ο πρόεδρος κύριος Τρισέ, δεν θεωρούμε ότι ο λέει λέει κ. Στοσέ, δεν θα πρέπει να, πάει, να πάει η Ελλάδα στο, στο, το να πάει η Ελλάδα στο, Ευρωπαϊκό, στο Διεθνές Ταμείο δεν το θεωρούμε πρόβλημα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι κάνει το Διεθνές Προσματικό Ταμείο. Τι κάνει, δύο πράγματα. Πρώτον, ορίζει και επιβάλλει πρόγραμμα προσαρμογής της οικονομίας μιας χώρας. Έχει ήδη γίνει αυτό. Τα ευρωπαϊκά θεσμικό όργανο το έχουν πράξει αυτό ήδη. Δύο φορέ χρειάστηκε να αναθεωρήσει η Ελλάδα στο αρχικό τη πρόγραμμα κατόπιν των πιέσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και το πρόβλημα που έχει τώρα η Ελλάδα δεν είναι διαφορετικό από αυτό. Μάλλον το πρόγραμμα που έχει τώρα η Ελλάδα δεν είναι διαφορετικό από αυτό που θα τη υπέδεικνυε το δουνού Δεν βλέπω δηλαδή προστιθέμενη αξία από μια προσφυγή στο Ιδρυτικό Ταμείο. Δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει το δουνού είναι να δανείσει χρήματα. Που όμω δεν θα αρκούσαν επουδενή να καλύψουν τις ε, ανάγκες Ελλάδας, είτε εφέτος του, του χρόνου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ρόλο μάλλον καταλητικό, δηλαδή επιβάλλει πρόγραμμα, δανείζει χρήματα και αναμένει ότι με το διτό αυτό του ρόλο μπορεί να ανακτήσει την οικονομική της δραστηριότητα μια χώρα για να βγει από την κρίση. Ε, αυτό πρέπει, μπορεί και πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το να πάει μια χώρα μέλος Τη ζώνη του ευρώ στο διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, το μόνο που βλέπω να έχει σαν συνέπεια θα ήταν να ερμηνευθεί σε επίπεδο διεθνέ ω μήνυμα αδυναμία των θεσμικών μα οργάνων ή του θεσμικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο θα ήταν ει βάρο ολόκληρης της Ένωσης, αν συνέβαινε. Και δεν βλέπω και την ανάγκη, αφού μπορούμε να το πράξουμε μόνοι μα. Γιατί να εμπλέξουμε άλλους οργανισμούς είναι σημαντικό να δώσουμε εμείς τις, επενδύ, απαντήσεις. Και επίσης η Ελλάδα δεν χρειάζεται σανίδα σωτηρίας. Έχει ένα πρόβλημα η Ελλάδα. Προσέφυγε στις αγορές, πλήρωσε πιο ακριβά την πίστοση, ναι, αλλά αυτό είναι ο κίνδυνος, ότι όταν κάνει τις θέση πληρώνει πιο υψηλό επιτόκιο. Είχε την πρόσφυγη στις αγορές και βραχυπρόθεσμα, εάν χρειάζεται υποστήριξη σε ρευστό μπορούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά απόψή μου να το προσφέρουν αλλά σαν είδα σωτηρίας δεν χρειάζεται γιατί θα εξακολουθήσει να αποπληρώνει το χρέος της και να πληρώνει τα επιτόκια όπως πρέπει για το χρέος της η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο από αυτό που έχει κάνει και το προσαρμοστικό, το νέο της πρόγραμμα δείχνει ότι έχει μπει στο σωστό δρόμο. Και το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαρκεί επίσης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Άλλο χρόνο δυστυχώς δεν έχω πλέον. Μέλο. Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω στα πορτογαλικά, που είναι επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Μιλάτε, μιλάω για το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, άρθρα 13 και 14. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εκδώσει συστάσεις και οδηγίες και να δώσει και τις ε, σχετικές ε, πληροφορίες. Τώρα, η BPN και η BPPS ε, αυτή τη στιγμή το ένα είναι εθνικοποιημένο και το άλλο είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα τα οποία έδωσε κάτω από, την, από το τραπέζι ε, και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γενικεύεται για ολόκληρη την Ευρώπη και δεν ε, το λέω αυτό για να επικρίνω την εθνική μας ε, εποπτεία, όχι κύριε Δικητά, αλλά η ερώτησή μου αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν, εφόσον συνέβη αυτό στην BPN και, και ακόμα και συμβαίνει και στην BPP, ξέρατε από το 2002 μέχρι σήμερα η Κεντρική Τράπεζα τι λένε αυτά τα, πρωτόκολλα, ε, αυτά τα άρθρα του πρωτοκόλου και τι ισχύει σε θέματα εποπτείας. Ζητήσατε πληροφορίες σε σχέση με την ε, μακροπροληπτική λειτουργία και την εποπτεία. Και έπειτα να σας ρωτήσω κύριε Δικητά πώς ερμηνεύετε εσείς αυτά τα άρθρα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, η συνθήκη είναι ξεκάθαρη. Λέει στη συνθήκη ότι μόνο οι νέε αποφάσει μόνο μια νέα απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να δώσει στην ΕΚΤ λειτουργεί, ε, ελεγκτικές, εποπτικές μάλλον λειτουργίες. Κανένα πρωτόκολλο δεν μπορεί να υπερέχει, υπερισχύει αυτού του άρθρου της συνθήκης. Αυτό που λέει είναι πως βέβαια η ΕΚΤΕ θα πρέπει να συνεργάζεται και να στηρίζει τον εποπτικό ρόλο στην Ευρώπη. Αλλά η ίδια η ΕΚΤΕ δεν έχει αρμοδιότητες εποπτικές. Δεν τις έχουν δοθεί. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τρισέ, απαντώντας σε ερωτήσεις σας, σας απάντησε το ίδιο. Ε, θέσατε την ίδια ακριβώ ερώτηση και είπε το ίδιο, πως η ΕΚΤ δεν έχει ευθύνη σε αυτόν τον τομέα, αυτό καθ' αυτό. Πρέπει να συνεργάζεται, να στηρίζει, αλλά δεν έχει αρμοδιότητα. Άρα λοιπόν και ο πρόεδρος Τρισέ απάντησε με τον ίδιο τρόπο και είπε πως δεν έτεθαν σχετικά ερωτήματα γιατί δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Και τώρα, για την εκτίμηση των καταθέσεων δεν είναι αλήθεια. Για στην περίπτωση της BPN, όπως γνωρίζετε, αυτό το οποίο διακυβεύεται στην BPP ε, δεν είναι οι καταθέσεις, είναι προϊόντα της ε, κεφαλαίου όπως ε, είχε προβλέψει και η εποπτική αρχή χρεοτήτλων και αυτά είναι τίτλοι, είναι προϊόντα, δεν είναι καταθέσεις. Ευχαριστώ. Αντολίνη Σάντζες Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κωνστάνσιο, εγώ εκτιμώ όλους ιδιαίτερος την πορεία σας και την επαγγελματική σας πείρα. Θέλουμε να βγούμε από την κρίση. Ο κύριος Τρισέ χτες είπε ότι ο πληθωρισμός δεν βρίσκεται στον ορίζοντα των προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τη γνώμη σας, πώς θα φροντίσει να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν κατάλληλες πιστώσεις για την ανάκαμψη. Πώς θα φροντίσουμε να μην υπάρξει πρόβλημα ρευστότητα, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να το πετύχει αυτό. Δεύτερον, δημοσιονομικά. Είναι γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις, να μην γίνει κάτι δυσανάλογο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν πώς θα συνεισφέρει ώστε να μην υπάρξει τέτοια δυσαναλογία. Τρίτον, όσον αφορά ε, τους οικονομικούς παράγοντες, πώς ε, θα μοιραστούν το βάρος που προκύπτει. Δεν πρέπει να ε, Υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις τράπεζες που πήραν βοήθεια και από αυτές που δεν πήραν βοήθεια. Και για το μέλλον υπάρξει μια συζήτηση. Μίλησατε για ένα ταμείο που θα βοηθούσε. Θα βοηθούσε ή θα διέλυε. Γιατί κινδυνεύουν οι αποταμιεύσει. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όπως είπα και πριν, το γεγονός ότι σήμερα προσπαθούμε και μειώνουμε κάπως τα προβλήματα που έχουν προκύψει και φροντίζουμε να δίνουμε ρευστό, δεν σημαίνει ότι κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Παρά τις αποφάσεις που πήραμε, μέχρι τώρα δεν υπήρξαν αλλαγές όσον αφορά τα επιτόκια. Δεν έχουν υπάρξει αλλαγέ εκεί εξαιτία των μέτρων που εμεί υιοθετήσαμε. Και όπω σου είπα και πριν, τα υιοθετήσαμε, αλλά δεν χρειάζονται πια. Τώρα λειτουργούν οι τράπεζες κανονικά, με ρευστό, έχουν όσο ρευστό τους χρειάζεται και δεν τους δημιουργήθηκαν δυσκολίες από τη στρατηγική που αποφασίσαμε αν υπάρχουν προβλήματα με την πιστοτική ικανότητα, αυτό δεν έχει να κάνει με την ρευστότητα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επί ευκαιρία, είναι αδύνατον να διακρίνουμε από την εξέλιξη των πιστώσεων τη ζήτηση η οποία έχει πέσει λόγω της ύφεση και τους περιορισμούς που έχουν εισαγάγει οι ίδιες οι τράπεζες. Όσον αφορά τώρα τα δημοσιονομικά των χωρών, όπως είπα, τα πακέτα που εγκρίθηκαν δεν ήταν πολύ μεγάλα, Οπότε νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη προοπτική σε όλα αυτά. Τα επιτόκια στις αγορές, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθορίζονται από την αγορά. Αν οι αγορές νιώθουν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικών εξαιτίας των ελλημάτων, μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα, κάτι το οποίο θα ήταν κακό για την ανάπτυξη και για την ανάκαμψη. Άρα υπάρχουν δύο πλευρές αυτό το νόμισμα. Άρα λοιπόν είμαστε στην οξία φάση της κρίσης. Την ξεπερνάμε και πια πρέπει να ζητήσουμε από τις χώρες να φροντίσουν για την εξυγίανση των δημοσιονομικών τους. Κάτι το οποίο μπορεί να έχει και θετικό αντίκτυπο στα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτόκια. Πολύ βασικό για την ανάκαμψη. Τέλος. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Οι εισφορές πρέπει να δοθούν από τις τράπεζες γενικά γιατί είναι όπως ο ρόλος που έπαιξαν πολλές ε, τράπεζες στην Αμερική με το FDIC. Στόχος δεν είναι η διάλυση. Εμείς θέλουμε αναδιάρθρωση και ενδεχομένως επαναπόλυση του οργανισμού, χωρίς όμως να τον διαλύσουμε. Και από την αρχή της κρίσης το FDIC ασχολήθηκε με πάνω από 400 τράπεζες στις Ηνωμένε Πολιτείε, ορισμένες από αυτές πολύ μεγάλες. Και αν τις συγκρίνουμε και με τις δικές μας τράπεζες. Και αυτό έγινε με ήπιο τρόπο. Ωραία, αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ξεχνάω το χρόνο κι εγώ. Παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντσιο, δώσατε μια εξαίρετη εικόνα για τα κριτήρια για μια καλή χώρα ενιανομίσματος, μια καλή περιοχή ενιανομίσματος. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η Καλιφόρνια. Δηλαδή η έλλειψη πολιτικής ένωσης δεν, δεν υπάρχει. Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα είναι αυτό που είναι, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι η εποπτεία πρέπει να είναι πολύ αυστηρή όταν έχουμε να κάνουμε με το σύμφωνο σταθερότητας και με την ε, εισδοχή σε αυτό. Οπότε εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό, δηλαδή τι θα σας ικανοποιούσε εσά, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό για την επιτυχία του ευρώ. Ο κύριος Κωνσταντσιο. Η Ελλάδα δεν είναι η Καλιφόρνια, εννοείται. Αλλά θέλω εδώ να σας υπενθυμίζω. Είπαμε και η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει δημοσιονομικά προβλήματα αλλά α πάμε στη Νέα Υόρκη πριν από μερικά χρόνια. Η Νέα Υόρκη επίση είχε πρόβλημα και η Ουάσιγκτον, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αρνήθηκε να βοηθήσει. Οπότε η Νέα Υόρκη έπρεπε να φροντίσει να κάνει τις δικές της μεταρρυθμίσεις, να υιοθετήσει τα δικά της μέτρα για να ε, ανακτήσει την αξιοπιστία της στις αγορές. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε μια νομισματική ένωση, που είναι και πολιτική ένωση, μπορεί να συμβεί με μια χώρα. Σα είπα, η κεντρική κυβέρνηση στην Αμερική, ο Άσιγκτον, δεν βοήθησε τη Νέα Υόρκη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που είναι αναγκαίο είναι μηχανισμοί που να διασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής πίεση πάνω σε μια χώρα μέλος, ώστε να πάρει τα μέτρα που πρέπει. Η δυσκολία στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ότι το πρόβλημα δεν εντοπίστηκε έγκαιρα από πριν. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Έτσι θα ήταν τα πράγματα πιο εύκολα για όλους και για την Ελλάδα ακόμα. Όμως τα μέσα υπάρχουν και μπορούμε να αναγκάσουμε τις χώρες να υιοθετήσουν τα μέτρα που πρέπει. Αν τώρα πρέπει να ενισχυθούν όσον αφορά το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας, θα έπρεπε ενδεχομένω ενδεχομένως, να φροντίσουμε για κάποιε κυρώσει. παρόλο που ορισμένε κυρώσει είναι δύσκολο να εφαρμιστούν. Άρα πρόληψη. Πρόληψη είναι αυτό που πρέπει να ενισχυθεί. Και αυτό το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας είναι που πρέπει να τηρείται. Και από εκεί και πέρα τα μέλη της ΟΝΕ, που αν μη τι άλλο έχουν ένα κοινό νόμισμα, οι χώρες λοιπόν, όλες οι χώρες πρέπει να καταλάβουν ότι, ότι όλοι κινδυνεύουμε να χάσουμε κάποια, κάποιο μέρος της κυριαρχίας μας όταν μπαίνουμε σε μία ε, νομισματική ένωση και όλοι πρέπει να το δεχτούν, να δεχτούν μεγαλύτερη ανάμιξη στις υποθέσεις τους προκειμένου να γίνονται προσαρμογές που επιβάλλονται. Όλα τα θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σε αυτό, να φροντίσουν να είναι έτσι τα πράγματα στο μέλλον και να μην έχουμε μια κατάσταση όπως είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πολύ αυστηρή εποπτεία. Αυτό είναι το αναγκαίο. Ευχαριστούμε. Τώρα, Άλντε, δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει ποιος θα πάρει τον λόγο. Όλετ Σμιτ. Ευχαριστώ. Επειδή έχουμε μεγάλη ισότητα μεταξύ μας, αποφασίζουμε τελευταία στιγμή. Κύριε Κωνστανσίου, Νομίζετε ότι το κύριο πρόβλημα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η κερδοσκοπία. Πρώτον. Και δεύτερον. Βεβαίω είστε ικανότατο οικονομολόγο, αλλά και πέραν αυτού, από τη γενική σα ε, εμπειρία στην ε, Κεντρική Τράπεζα και από τα όσα ακούσαμε και τον Ιανουάριο και τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει μια διαφανή αγορά με καλύτερη επιτήρηση και πρέπει αυτή να υπάρχει ή θα έπρεπε κάποια στοιχεία να διαγραφούν, κάποια προϊόντα να διαγραφούν, να απαγορευτούν ορισμένα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων. CDF, CDS, βραχυπρόθεσμος, υπολογισμός κτλ. Ο κύριος Ζωνκλώτ Κρισέ αλλά και άλλοι χτες ήταν ε, πιο προσεκτική. Εγώ προσωπικώς ως φιλελεύθερος δεν είμαι τόσο υπέρ της απαγόρευσης των συγκεκριμένων προϊόντων, γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιο προϊόν που θα θέλουμε να απαγορεύσουμε. Απάντηση. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Να σας πω, το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μόνο κερδοσκοπία, σε μεγάλο βαθμό ναι, αλλά αλλά ακόμη και η ασφάλιση θέτης πληρωμών ε, είναι, έχει πολύ μικρό περιθώριο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να επηρεάσει δηλαδή ουσιαστικά το spread ε, το οποίο καταβάλει στην αγορά το, τη χρηματοπιστωτική ίδια η κυβέρνηση. Δεν είναι, ζήτημα λοιπόν ε, μόνο κερδοσκοπίας. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απαγόρευσης ορισμένων προϊόντων. Αυτό που είπα στην παρέμβασή μου είναι ότι ιδιαίτερα αυτά τα CDS θα πρέπει να προχωρούν προς μια οργανωμένη ε, αγορά, χρηματιστηριακή αγορά, οργανωμένη αγορά. Αυτό θέλω να γίνεται και θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά η δυνατότητα της ε, πώλησης καθαρά βραχυπρόθεσμων πωλήσεων των CDS, μόνο, μόνο των υποθέσεων, δηλαδή αθέτησης πληρωμών. Μόνο και μόνο γιατί αυτά τα μέσα έχουν ρόλο ασφαλιστικό καταρχάς και όχι άλλον. Δεν πρέπει να πολλούνται γυμνά δηλαδή. Όπως θα σας πει οποιοδήποτε οικονομολόγος που έχει μελετήσει αυτήν την κρίση, η πώλησή τους γυμνή, σκέτη, έχει γίνει καταχρηστικά και κερδοσκοπικά μόνο. Σε ένα μέρος λοιπόν η κρίση, σε ένα μέρος η αποτυχία ορισμένων θεσμών έχει να κάνει με τον ρόλο αυτών των ε, ασφαλίστρων. Έχει καταστρατηγηθεί η αρχική τους, ε, ο αρχικός του σχεδιασμός, καταχρηστικά χρησιμοποιούνται όπως είπα και θα πρέπει ίσως η πώλησή τους, η βραχυπρόθεσμη γυμνή πώλησή του, η ε, υψηλή πώλησή του αν θέλετε, να απαγορευτεί. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα θα ήθελα ήμουν υπέρ μια οργανωμένη χρηματοπιστωτική αγορά ρυθμιζόμενη. Κάποιοι από τους ε, οικονομολόγους πάλι για την ε, απαγόρευση της ψηλής βραχυπρόθεσμης πώλησης αυτών των CDS έχουν ακόμη και υποστηρίξει την ιδέα αυτή, αν και εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, απόλυτης απαγόρευσης τους, γιατί θα οδηγούσε την αγορά σε αδράνεια. Ο πολιτής που πουλάει ένα CDS σε κάποιον που έχει συμφέρον ασφαλιστικό, θα πρέπει από αλλού να καλυφθεί, να αντασφαλιστεί Και άρα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα έστω και μόνο το ασφάλιστρο να αγοραστεί. Άρα όχι πλήρη και απόλυτη απαγόρευση. Αυτό θέλω να πω. Για τον τεχνικό αυτό λόγο, για τη δυνατότητα της ατασφάλισης δηλαδή. Αυτό για να διευκρινίσουμε τις απόψεις μου. Όπως βλέπετε δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ από το όσα είπε ο διοικητής Δράγκη και ο διοικητής Τρισέ. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία Κούνη. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Κωνσταντσιο, οι συνθήκε, διαπίστωσαν ότι δεν επιτρέπουν την έκδοση ευρωομολόγων σήμερα. Όμω, ας υποθέσουμε, υποθέσουμε ότι αλλάζει, αλλάζουν οι συνθήκες και μπορούμε να εκδώσουμε ευρωομόλογα. Εσείς πώς αναλύετε μια τέτοια προπτική έκδοση σε ευρωομολόγων. Θεωρώ ότι τα ευρωομόλογα μπορούν να εγγραφούν σε μια συντονισμένη στρατηγική σαν ένα μέσο που βοηθάει τις χώρες να είναι πιο ανταγωνιστικές. Ίσως έτσι να μπορούμε να παρεύουμε καλύτερα σε περιπτώσεις κρίσεων όπως η σημερινή. Δεν θέλω να μου πείτε τι πιθανότητες βλέπετε η, η Ευρώπη να έχει τέτοια ευρωμόλογα, αλλά πιστεύετε εσείς ότι θα βοηθούσανε. Νομίζω ότι έχω ήδη απαντήσει την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ σε αυτή την ερώτηση. Δεν νομίζω ότι τα ευρωομόλογα μπορούν να εκδοθούν για να αντικαταστήσουν το χρέος μιας χώρας μέλους, δεν θα έπρεπε να αποτελούν μέσο για να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνες, χρέη μιας χώρας μέλους. Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 123 η χρήση ευρωομολόγων προκειμένου να αντικαταστήσουν ή για να λύσουν ή για να μειώσουν ένα πρόβλημα χρέους κάποιας χώρας δεν είναι κάτι που συστήνω. Όμως είπα και την προηγούμενη φορά ότι αν σκεφτούμε προγράμματα επενδυτικά, ευρωπαϊκά, που να μπορούν να ενισχύσουν χώρες μέλη γενικά με δαπάνες στις υποδομές. Αυτό θα ήταν ένα πρόγραμμα που δεν θα είχε να κάνει άμεσα τίποτα να κάνει με το χρέος μιας χώρας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό και αυτό, είπα, μπορούμε να το σκεφτούμε. Δεν θα ήμουν αντίθετος στη χρήση τέτοιων μέσων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκδίδει ομόλογα για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες της ε, δικές της, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιου είδους προγράμματα θα μπορούσαν να ενισχυθούν σε περιόδους κρίσης. Από οικονομική δηλαδή άποψη δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να το κάνουμε. Αυτό ναι. Αλλά μην συγχαίουμε με το σημερινό πρόβλημα κρίσης εξαιτίας υπερβολικού χρέους χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Η υπερβάνωση πέρασε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δικητά, ε, κύριε Δικητά της Πορτογαλικής Εθνικής Τράπεζας λέει στη δεύτερη παράγραφο ότι και τα ε, λέει λοιπόν εκεί κάτι το άρθρο, το γνωρίζετε νομίζω και πιστεύω πως το χρειαζόμαστε όταν ε, ερμηνεύουμε το 123. Τώρα, όσον αφορά τα CDS, τις ασφαλίσεις καταθέτησης πληρωμών, δεν ήσασταν κατά απαγάρευσης ε, των ΣΕΝΤΕΕΣ που πολλούνται αφαιρέγγια ή χωρίς κάλυψη. Μα οι πολίτες δεν είναι ηλίθιοι, δεν καταλαβαίνουν γιατί στον τομέα των τροφίμων, στον τομέα της οδικής ασφάλειας παντού υπάρχουν ε, κείμενα για την τοξικότητα και έλεγχη για την τοξικότητα ή όχι των προϊόντων και τη δυνατότητα να αποσυρθούν από την αγορά από τη στιγμή που αποδεικνύονται ε, τοξικά. Γιατί λοιπόν και στον τομέα της οικονομίας να μην το σκεφτούμε λίγο αυτό. Και έπειτα, στην ατζέντα σα, εντάξει, είναι φορτωμένη και εξαντλητική. Αλλά βάζετε τέσσερι από τι. δέκα μάλλον από τέσσερι προτάσει. Μία από τι μεγάλε δυσκολίε που έχουμε όμω είναι ότι όλα αυτά ε, γίνονται μέσα σε μη συγκοινωνώντα αγκία και από τα όσα αναφέρατε για το θέμα το πώς θα προσανατολιστεί εκ νέου ο, η, ρύθμιση των αγορών ε, ώστε να συμβαδίζει με την πραγματική οικονομία μέσα σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και με τους επενδυτές δεν προβλέπεται. Εγώ δεν θέλω να επικρίνω την Επιτροπή της Βασιλείας που δεν το έκανε, γιατί δεν ήταν ο ρόλος της, αλλά τελικά είναι μια νομοθεσία την οποία έχουν εμπιστευτεί, έχουν μάλλον εμπνευστεί οι κεντρικοί τραπεζίτες μέσα στην Επιτροπή της Βασιλείας, ενώ δεν έχει γίνει δημοκρατικός διάλογος και συζήτηση. Εσείς ως κεντρικός τραπεζίτης αισθάνεστε ότι θα πρέπει να εμπλακείτε περισσότερο και έπειτα. Ο ίσως μελλοντικός σας πρόεδρος, ο κύριος Ζανκλώτ Τρισέ, μας λέει ότι ναι, ότι όλα αυτά είναι προς το συμφέρον της αμερικανικής οικονομίας. Ποιο συμπέρασμα εσείς ε, βγάζετε για την ε, πολιτική ε, συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ να εξηγήσω, γιατί το έχω πει 6-7 λεπτα έχουμε ακόμα για να ολοκληρώσουμε. θα μπορούσατε να έχετε κάνει και άλλες ερωτήσεις. Αν μου επιτρέπετε θα σας απαντήσω στα αγγλικά γιατί όπως σας είπα είμαι πιο ακριβής στη γλώσσα αυτή. Τα γαλλικά μου είναι λίγο σκουριασμένα. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και προηγούμενη έγκριση των προϊόντων αυτών, γιατί σε αυτό αναφερόσασταν, δεν πιστεύω πως είναι δυνατόν ή σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, αν, βάλουμε, αν δούμε τα CDS, την ε, την ασφάλιση για θέτηση πληρωμών. Όταν φτιάχτηκαν όλα αυτά, ήταν καλή ιδέα. Κανένας δεν μπορούσε να έχει προβλέψει στην αρχή το είδος της χρήσης που τους έγινε αργότερα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι χημεία ώστε να γνωρίζουμε αν είναι ή όχι κάτι τοξικό. Είναι κάτι πολύ πιο βέβαιο. Πάντως, Η προηγούμενη έγκριση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεν ξέρω αν είναι αυτό λοιπόν σκόπιμο. Αυτό που είναι απαραίτητο, όπως προτείνω μαζί με άλλους, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου σκέψεων. Δεν μπορείτε να βρείτε κανέναν ε, ε, ε, πιο, πιο φιλελεύθερο. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να, να, να σκοτωθεί, όπως λέμε, να εξαλειφθεί η σημερινή αγορά CDS. Και μετά να μετακινηθούμε σε μια νέα. Ναι. Αφού είδαμε λοιπόν πως κάποιος συμπεριφέρεται με λάθος τρόπο, θα έπρεπε να το έχουμε προβλέψει. Αυτή η αγορά είχε τελείως ξεπεράσει την κατάσταση, είχε φτάσει στα 62, 3 εκατομμύρια στην αιχμή της. Ορισμένες φάσεις αυτής της διαδικασίας που ήταν πολύ γρήγορη, η ΦΕΔ της Νέας Υόρκης έκανε, ε, κατέστησε δημόσια γνωστό πως ακόμα και οι υπολογισμοί, οι λογαριασμοί μέσα στους οργανισμούς αυτούς δεν γίνονταν σωστά γιατί δεν είχαν το χρόνο να επεξεργαστούν όλες αυτές τις συναλλαγές και ούτω καθεξής. Εκεί θα έπρεπε να έχει γίνει παρέμβαση προηγουμένως, όταν ήταν σαφές πως υπήρχαν προβλήματα. Γιατί αυτά τα μέσα, αυτά τα CDS, γιατί είναι, είναι μέσα μαζικής καταστροφής. Μια κέρια λοιπόν παρέμβαση στην κατάλληλη στιγμή είναι απαραίτητη, αλλά όχι προηγούμενη έγκριση προϊόντων, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί εκ των προτέρων να αναλύσει πώ θα λειτουργήσουν ή πώ θα γίνει η κατάχρηση αυτών. Και φυσικά πολύ αυστηρή παρακολούθηση τη κατάσταση. Όσον αφορά τώρα τα όσα προετοιμάζονται σε διάφορο πλαίσια και αναφέρονται και στον κατάλογο κτλ. Εσείς επικρίνατε την έλλειψη διαλόγου και ούτω καθεξής. Πρώτον, τη σήμερα μέρα τα πάντα είναι σχεδόν ε, διαφανή. Μπορεί κανείς να πάρει όλα τα έγγραφα, τις συζητήσει και όλα αυτά που γίνονται. Και η Επιτροπή της Βασιλείας ε, δεν έχει κάνει σφάλμα. Ό,τι και αν κάνει, και κάνει καταλήξει μάλλον η Επιτροπή της Βασιλείας, θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις διάφορες χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δημοκρατικά τη θεσμικά όργανα και το πλαίσιο το οποίο έχουμε και τον τόσο το οποίο λειτουργούμε. Εργάζεται λοιπόν σε τεχνικό επίπεδο και κάνει προτάσεις. Και έπειτα πρέπει να προετοιμαστεί η σχετική νομοθεσία και μπορεί να είναι διαφορετική. Ξέρετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τις δικές του αρμοδιότητες να συμμετέχει στη διαδικασία μετατροπής των προτάσεων σε νομοθεσία. Όσον αφορά την πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών, ξέρετε ότι για μεγάλες χώρες και μεγάλους οικονομικούς, ε, οικονομικές περιοχές όπως η Ευρωζώνη, το καθεστώς για την συναλλαγματική ισοτιμία είναι κειμενόμενο. Έχουμε ένα κειμενόμενο νόμισμα. Δεν υπάρχει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Δεν υπάρχουν ε, κλίμακες ανώτατα όρια ή οτιδήποτε. Ζούμε μέσα σε ένα καθεστώς κειμενόμενο κειμενόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και είναι και σωστό για μεγάλες ζώνες όπως η Ευρωζώνη. Άρα κειμενομενη συναλλαγματικη ισοτιμια και υπάρχουν για μεγάλε ζώνε μικρά, λίγα μέσα για να ασκήσει